Eh, να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη σημερινή μας συνεδρίαση. Να καλημερίσω όλους τους παρόντες, ολιγάριθμους προς τον παρόν, αλλά ελπίζω να γεμίσει η σιγα σιγά-σιγά. Είναι μικρή η Επιτροπή μας, ε, η Επιτροπή Αλίας, κύριε, κύριε Υπουργέ. Λίγοι αλλά καλοί είμαστε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Είχαμε με τον Υπουργό, οι Πρόεδρος και οι συντονιστές ε, προηγουμένως μια συνάντηση όπου συζητήσαμε ήδη κάποια από τα σημαντικά θέματα που θα αποτελέσουν και αντικείμενο της Πολωνικής Προεδρίας. Θα σας καλωσορίσω λοιπόν στην Επιτροπή Αλίας κύριε Υπουργέ. Σας έχω ήδη ευχηθεί κάθε επιτυχία για το εξάμεινο της Πολωνικής Προεδρίας στο πλαίσιο της εντολής που έχετε ως ε, Προεδρεύον του Συμβουλίου. Είναι μια αξιομνημόνευτη μέρα σήμερα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τι προτάσεις ε, για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής σήμερα. Είναι 13 του μήνα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τους Ισπανούς αυτός ο αριθμός, αλλά τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ ε, σημαντική μέρα για όλους μας αυτή. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πρόσφατα επισκέφθηκε την Πολωνία μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σας και πάντοτε έχετε δείξει προθυμία να συνομιλείτε με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διπλά σας ευχαριστώ λοιπόν και για την ε, ε, διαθεσιμότητά σας ε, να συνεργάζεστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό λέει πολλά υπέρ σας. Και σίγουρα θα είναι ευεργετικό και για τις ε, μελλοντικές μας σχέσεις, ιδίως στα θέματα της συναπόφασης ή της κανονικής, ε, της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα σας δώσω το λόγο για να εξηγήσετε στους συναδέλφους μας ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Εν συνεχεία θα περάσουμε σε ένα γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων εφόσον το επιθυμούν ή θα δώσω το λόγο σε οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο επιθυμεί. Νομίζω ότι είναι καλό οι συντονιστές εδώ δημοσία να εκφράσουν τις απόψεις των πολιτικών ομάδων και να δώσουμε τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους συναδέλφους της Επιτροπής μας να διατυπώσουν και αυτοί τα ερωτήματά τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Υπουργέ, σας δίνω το λόγο. Przewodnicząca, Panie i Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τι προτεραιότητε τη Πολωνική Προεδρία. Δεν πειράζει που δεν είναι πολλοί παρευρισκόμενοι οι βουλευτέ. Έχω μακρά πολιτική εμπειρία και πολλέ φορέ έχω μιλήσει σε αίθουσε που μπορώ να σα πω δεν είχε σχεδόν καθόλου παρευρισκομένους εκτός από τους ομιλούντες. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στον κοινοβουλευτισμό. Δεν είμαι προληπτικό εξάλλου και δεν με πειράζει καθόλου που είναι 13 του μηνό σήμερα. Στην Πολωνία έχουμε καλέ εμπειρίε με τη 13η, γιατί στι 13 Δεκεμβρίου του 1980 ξεκίνησε η πτωτική πορεία του κομμουνιστικού καθεστώτος και το 2002 η ίδια ημερομηνία ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, μάλλον ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το 13 του μηνός δεν είναι καθόλου αρνητική, ε, αρνητική ημερομηνία. Θα έλεγα ότι είναι και τυχερή μας ημερομηνία. Περνώ όμως ε, στα σημερινά μας θέματα. Κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα, διότι αναλαμβάνει η Πολωνία την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω εγώ την τιμή να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της αλληλευτικής πολιτικής ε, για την Προεδρία μας. Για την Πολωνική Προεδρία, αλλά και για μένα προσωπικά, είναι σημαντική επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή Αλίας ιδίω όσον αφορά το νομοθετικό έργο στον τομέα της αλίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία που θα έχουμε κατά το εξάμεινο αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε πολλά θέματα. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου, τον Προεδρεύοντα της Ουγγρικής Προεδρίας, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Η Ουγγρική Προεδρία κατόρθωσε να ολοκληρώσει δύο σημαντικά θέματα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Διεξήχθησαν και πολλοί επικοδομητικές συζητήσεις και για τη μεταρρύθμιση της ε, αλίας και για τα δικαιώματα και για τις ποσοστώσεις της αλίας το 2012 και άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω ότι και η Πολωνική Προεδρία θα μπορέσει να συνεχίσει με επιτυχία τις αντίστοιχες συζητήσεις. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, προγραμματίζουμε συζήτηση των θεμάτων ε, αλία στο Συμβούλιο τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, μπορεί να προκύψουν ε, και άλλες συζητήσεις για θέματα αλίας. Οι πιο σημαντικέ προτεραιότητε για τον τομέα τη αλλία κατά του επόμενου μήνε είναι οι εξή. Πρώτον, μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική καθορισμός των ΤΑΚ και των ποσοστώσεων για το 2012, καθώς και σχέδια οικονομικής διαχείρισης. Θα περάσω τώρα στα θέματα αυτά λεπτομερώς. Το φθινόπωρο θα γίνουν οι συζητήσεις για την νομοθετική πρόταση για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσει αυτές, αλλά πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία ήδη έχει ξεκινήσει, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο απόφασης των σχετικών ε, μέτρων και την επόμενη Τρίτη θα συζητηθεί στο Συμβούλιο το θέμα αυτό και θα δούμε και τις ε, τεχνικές συζητήσεις ε, που θα γίνουν για θέματα λεπτομέρειας. Ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση για όλα αυτά. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση για το βασικό κανονισμό και συζητείται και η κοινή οργάνωση της αγοράς παράλληλα γίνεται μια συζήτηση μεταξύ Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου, μεταξύ ε, των ε, τριών χωρών για την Προεδρία και ε, υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των συμφερόντων του, του τομέα της αλίας. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Προεδρία μας θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει συνέχεια και συνέπεια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για το περιεχόμενο της κοινή πολιτικής αλληλείας. Αυτό θα το κάνει η Επίτροπος. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να μιλήσουμε για τους μηχανισμούς της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, που είναι σωστοί μηχανισμοί. Επίσης, ένα ιδιαίτερο θέμα ενδιαφέροντος είναι η ηχθειοκαλλιέργεια, που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 21ο αιώνα. Ένα σημαντικό τμήμα της μεταρρύθμισης είναι και η χρηματοδότηση του τομέα από ε, αυτό που θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας. Το Νοέμβριο θα έχουμε πρόταση της Επιτροπής ε, και περιμένουμε ε, τις προτάσεις και την ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Η λεπτομερής εξέταση αυτών των θεμάτων θα γίνει στη συνέχεια από τη Δανική Προεδρία. Περνώ τώρα στη δεύτερη προτεραιότητά μου για τις αλληλευτικές δυνατότητες κατά το 2012. Υπάρχουν τέσσερα βασικά ζητήματα. Πρώτον, μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με τον σωστό τρόπο. Δεύτερον, αλληλευτικά αποθέματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Κάτι που δεν είναι απλό, αλλά πλησιάζει η τελική ημερομηνία του 2015 που έχουμε θέσει και δεν μπορούμε να αφήσουμε την προθεσμία αυτή να πάει χαμένη. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε τα αλληλευτικά αποθέματα και να μην αφήσουμε κανένα είδος ε, να καταστραφεί. Είναι κάτι ε, στο οποίο έχουμε δώσει προτεραιότητα και θέλουμε να συνεχίσουμε. Το πιο δύσκολο πρόβλημα νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων. Η Επιτροπή προτείνει διάφορες μεθόδους. Προτείνει έναν υπολογισμό ε, της μείωσης κατά 25% του αποθέματος και καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι. Γι' αυτό ένα σοβαρό θέμα για το Συμβούλιο είναι η έλλειψη των ε, σωστών επιστημονικών δεδομένων και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. τα σχέδια οικονομικής διαχείρισης ε, είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Τίθενται μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, με βιώσιμο τρόπο τα αλληλευτικά αποθέματα προς όφελος και των αλλιέων το αδιέξοδο στο οποίο έφτασε η ε, θεσμική πολιτική, ιδίως όσον αφορά ε, το σκουμπρί και ε, άλλα είδη, είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν και θα θέλαμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σωστή συμβιβαστική λύση. Για τα σχέδια μακροπρόθεσμης διαχείρισης, το σχέδιο για τον ερυθρό τόνο ε, είναι επίσης μία από τις προτεραιότητές μας και το τωρινό ε, πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί από την ε, ΙΚΑΤ, από την Διεθνή Επιτροπή Διαχείρισης των Νοηδών. Συζητήσεις γίνονται και με την Νορβηγία και αυτό έχει σχέση με το σκουμπρί που σας προανέφερα και ελπίζουμε ότι θα επιτευχθούν πρόοδοι και με την Ισλανδία και με τις νήσους Φερόες. Ε, χρειαζόμαστε μια κοινή ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε ε, να καθορίσουμε αποδεκτά, αποδεκτές ποσοστώσεις για όλες αυτές τις χώρες. Ελπίζουμε ότι η ετήσια συνάντηση της ΙΚΑΤ ε, θα αντιμετωπίσει λιγότερα αντιφατικά θέματα από ό,τι πέρυσι, γιατί υπήρχαν ε, αρκετές συγκρούσεις στην ε, Επιτροπή κατά την προηγούμενη χρονιά. Στον τομέα της αλληλείας υπάρχουν και σημαντικοί τομείς εταιρικής σχέσης που θα ήθελα να αναφέρω και εδώ έχουμε τη συνεργασία με την εταιρική σχέση με τη Μαυριτανία, με την Γρυλανδία και το Μαρόκο. Για το Μαρόκο ε, παρατείνεται κατά ένα έτος η αντίστοιχη συμφωνία και ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκριση για την ε, παράταση της συμφωνίας. Ε, είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχουν πολλές πολιτικές παράμετροι. Θέλουμε και ο τοπικός πληθυσμός να υποφελείται από τις συμφωνίες αυτές και να έχουμε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη ε, συμφωνία και εταιρική σχέση. Οι τελευταίοι 18 μήνες, κύριε Πρόεδρε, έδειξαν ε, πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα της αλίας. Ο στόχος μας είναι να έχουμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρώπης. Πάντοτε υπάρχουν διαστάσεις απόψεων και το σημαντικό είναι εμείς ως πολιτικοί να αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ακούμε αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες και να μπορούμε να βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις. Η Πολωνική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει τον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο κατάλληλος τρόπος για να επιτύχουμε φιλόδοξα ε, προγράμματα, όπως ε, το δικό μας ε, κατά το επόμενο εξάμεινο της Πολωνικής Προεδρίας. Τονίζω για άλλη μια φορά ότι για μας είναι πολύ σημαντική η καλή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τακτικές συζητήσεις, όπως η σημερινή συνάντηση, για να μπορούμε εγκαίρως να ενημερωνόμαστε για τις αποφάσεις των υπολείπων θεσμικών οργάνων και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σωστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ εκ νέου για την πρόσκληση που απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο καταρχάς στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και εν συνεχεία στους υπόλοιπους βουλευτές της Επιτροπής μας. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο λοιπόν με τους συντονιστές και δεύτερο με τους υπόλοιπους ομιλητές. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, η κυρία Πατάνιβιτς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μία ακόμη φορά καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να αναφερθώ στην έξοχη δουλειά, στην έξοχη προετοιμασία που κάνατε όσον αφορά την έναρξη του διαλόγου με το Κοινοβούλιο, ένα έναρξη ενός ευρέως διαλόγου αναφέρω ο υπουργό το ότι σε κάποιες φάσεις δεν θα μπορέσουμε να ε, συνάψουμε, να συνάπτουμε συμφωνίες που καλύπτουν τα πάντα. Αλλά μάλλον να, έχουμε, να συμφωνούμε σε όλα, αλλά είναι καλό να έχουμε τακτικό διάλογο το Κοινοβούλιο με την Προεδρία και έτσι θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Εφόσον έχω το λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ στην παρούσα κατάσταση. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής να είναι μια γενική μεταρρύθμιση ούτως ώστε να εξαλείψει τα προβλήματα που δεν έχουν ικανοποιηθεί ε, ικανοποιητικά. Εν γέννη, όσον αφορά αυτά που θα παρουσιαστούν το απόγευμα, δεν θέλω να προβλέψω ή να προδικάσω, αλλά αυτό που θα λάβουμε σαν πρόταση θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του ελευτικού τομέα, τις προσδοκίες επίσης του Κοινοβουλίου. Υπήρχε γενική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτρόπου όταν συζητήθηκε η πράσινη βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή αληθικής πολιτικής. Με βάση όλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό. Τι είδους μέτρα θα λάβετε ούτω ώστε πραγματικά να εφαρμοστούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα θέσετε σάρκα επί των οστών που αποτελούν τα διάφορα θέματα για την μεταρρύθμιση. Η περιφερειοποίηση, παραδείγματο χάρη, αυτό είναι κάτι που ήδη αναφέρθηκε, διάφορα ε, μοντέλα διαχείρισης. Ε, τι θα γίνει με τις στρατηγικές. Στρατηγικές για την καταπολέμηση ε, των απορρίψεων και των παρανόμως αλληλευωμένων ηχθείων. Μία άλλη πτυχή που ανέφερα στο πρωινό. Ε, η επιστημονική βάση για τη λήψη αποφάσεων για τα ΤΑΚ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πολιτικές αυτές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται επί επιστημονικής βάσεως. Το ζήτημα είναι πόσο αξιόπιστες θα είναι οι μελέτες οι οποίες επηρεάζουν τον τομέα σε κάποιες περιφέρειες μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει ανάγκη μιας προσπάθειας να κινηθούμε προς μια γενική βάση που θα ε, αποφαίνεται επί της αξιοπιστίας των επιστημονικών ερευνών. Όταν συντάσσονται για κάποιες χώρες ή για κάποιους τομείς αυτές οι εκθέσεις, ε, δεν υπάρχει, δεν αντιμετωπίζονται με μεγάλη αξιοπιστία. Γιατί και οι χώρε προσπαθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά του. Υπάρχουν και διάφορα τεωμεακά προβλήματα. Η μονομερής απόφαση της Ισλανδίας για την δημιουργία, για τη θέσπιση ποσοστώσεων είναι κάτι που μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τρίτες χώρες με τρίτες χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε ε, την αλία διαφόρων αποθεμάτων. Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει σωστή πρακτική στον αφορά την αλληλεία, ενώ ακολουθούμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση σωστή πρακτική. Άρα πρέπει να έχουμε εμείς μια θέση εναντί αυτών των χωρών. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσω συμφωνιών. Γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων αυτές τι συμφωνίες. Πολύ συχνά μας παρουσιάζονται τελεσμένα γεγονότα και πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Δεν ε, πρέπει να αναγνωριστεί ότι είμαστε κοινοβούλιο εδώ. Και σαν κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει να επιληθούν τα αλληλευτικά προβλήματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ Υπουργέ. Σας ευχαριστώ Ρόντου, από την ομάδα Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω ε, στην Επιτροπή μας και χαίρομαι που θα μας δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά και ε, ήδη μετά από τη σημερινή πρωινή μας συνάντηση κατά το πρωινό και ότι θα είναι πολύ επικοδομητική η συνεργασία μας. Πρέπει να δούμε την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια μεταρρύθμιση η οποία είναι σημαντική. η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο θα πρέπει να συναποφασίζουν και αυτή η ευθύνη θα πρέπει να μας οδηγήσει στα ορθά αποτελέσματα. Η παλαιά μεταρρύθμιση ήταν πραγματική πολιτική καταστροφή. Θέλουμε να αποφύγουμε την υπεραλίευση, θέλουμε να αποφύγουμε ε, τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα σε μεγάλο βαθμό και να αποφύγουμε και τις συνεχείς παραβιάσεις στο πλαίσιο της παράνομης και άναρχης αλίας. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία και αποδοχή των απόψεων μεταξύ αλλιέων, επιστημόνων και πολιτικών. Είμαι πεπισμένη ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε ε, το καθήκον μας και να έχουμε βιώσιμη αλία. Ε, χρειαζόμαστε μια ε, επάνωδο των περιφερειακό χαρακτήρα της αλίας. Δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες σε όλες τις περιοχές ε, με βάση τα προβλήματα κάθε περιοχής. Και ξέρω ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα από αυτού. Και το είπαμε εξάλλου και στην Επίτροπο σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις. Χρειαζόμαστε επιστημονικά δεδομένα και έρευνα για νέα αλλιευτικά εργαλεία και δεν χρειαζόμαστε επιδοτήσεις που θα επιβραβεύουν την παράνομη και άναρχη αλληλεία. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ταμείο για την αλληλεία, διότι χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Χρειαζόμαστε ελέγχους συνεπείς και ε, θα πρέπει να ανελαμβάνουν την ευθύνη τους και οι ελεγκτικές αρχές και οι αλληλείς. Το 40% των αναγκών μας το προμηθευόμαστε από την Αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 60% από χώρες εταίρους. Και γι' αυτό είναι εύλογο το ότι πρέπει να συζητάμε τα θέματα των αλλιευτικών συμφωνιών και των εταιρικών σχέσεων. Χρειαζόμαστε αυτές τις εταιρικές σχέσεις. Και όταν λέμε ε, εταιρικές σχέσεις δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όσον αφορά τον προπολογισμό, το Συμβούλιο προτείνει μια μείωση 6,8% και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Υπουργέ ήδη από αυτόν τον πρώτο γύρο ε, να μας εξηγήσετε ε, πώς έχει η κατάσταση σχετικά με τις μειώσεις του προϋπολογισμού. Θα ήθελα ήδη από τώρα στην απάντησή σας να μας πείτε ότι είστε κατά αυτών των περικοπών για την αλληλεία, γιατί αυτό θα δώσει ένα σημαντικό θετικό σήμα για τη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ο κύριος Υπουργό είναι εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας εδώ. Δεν έχει έρθει από την ιδιότητα του, υπουργού, ε, του Πολωνού Υπουργού, ο ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω όπως οι συνάδελφοί μου τον Υπουργό είτε υπό την ιδιότητα του Πολωνού Υπουργού είτε του Προεδρεύοντο τη Πολωνική Προεδρία και να του εκφράσω κάθε επιτυχία για το εξάμεινο τη Προεδρία. Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που προσφέρθηκε να μα συναντήσει πριν τη συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Σέβομαι βέβαια. Ε, μάλλον θα ήθελα να προτείνω ίσως μετά τις ε, συνεδριάσεις ε, του Συμβουλίου να συναντηθούμε. Τώρα το Δεκέμβριο είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τον Οκτώβριο εντάξει, ίσως καλύτερα θα ήταν πάντως να μας ενημερώσει μετά και όχι από τον προτέρα να συναντηθούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τα ψάρια και τα λευτικά προϊόντα, σίγουρα υπάρχει το θέμα της πληροφόρησης ε, των καταναλωτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο Κοινοβούλιο και ιδίως για τη δική μας πολιτική ομάδα. Η Προεδρία σας πώς ε, προτίθεται να προωθεί τον κώδικα διοντολογίας του ΦΑΟ για υπεύθυνη αλία καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές ε, του ΦΑΟ για την οικολογική σήμανση των ε, ψαριών και των αλληλευτικών προϊόντων. Σήμερα, κατά σύμπτωση, είναι η μέρα που ε, παρουσίασε η Κομισιόν τις προτάσεις της για την κοινή αλληλευτική πολιτική και βέβαια ελπίζουμε να είναι σε βάθος αυτές οι προτάσεις ούτως ώστε να επιτραπεί η εκβάθρον μεταρρύθμιση η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη ίσως να μην είναι τόσο ριζική όσο εμείς θα την επιθυμούσαμε αλλά τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα εδώ στο Κοινοβούλιο χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, να την επεξεργαστούμε την πρόταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν πολλές φορές ε, μας έχει πει ότι είναι υπέρ της περιφερειοποίησης. Σήμερα με εξέπληξε αυτό που είπατε κύριε Υπουργέ για την βαλτική και την περιφερειοποίηση. Είπατε ότι δεν μπορούμε με ένα μέγεθος να τα καλύψουμε όλα. Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική μεταρρύθμιση και η περιφερειοποίηση θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική ε, διαδικασία ε, διαχείρισης για να έχουμε αποτελεσματικότητα, να έχουμε φθηνές τιμές και να υπάρχουν τοπικές ε, δομές διαχείρισης που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν άμεσα τα ζητήματα. Και πριν προλάβει να πει κανεί ότι μιλάμε για επανεθνικοποίηση, δεν πρόκειται περί αυτού. Ουσιαστικά επιδεικνύουμε ρεαλισμό. Εσείς ίσως είστε, είστε πιο εξοικειωμένο ε, ή θα είστε πιο εξοικειωμένο με κάποιες νομικές πτυχές. Μπορεί κάποιος να πει αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ε, νομίζω όμως ότι αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή πολιτική βούληση και ιδίως από εσάς κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου στη διάρκεια του εξαμήνου σας. Για τις ε, απορρίψεις δεν νομίζω ότι αρκεί να πούμε ότι πρέπει ε, να σταματήσει η μάστιγα αυτή ε, και να σταματήσουν οι απορρίψεις. Αλλά ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας ε, δώσω εγώ συμβούλια. συμβουλίες, κύριε Πρεδρεύοντα. Οποιοςδήποτε επίτροπος ή πρόεδρος λέει ότι θα έχουμε μηδενική πολιτική απορρίψεων. Θα αποτύχει αυτός που θα το πει αυτό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να το αντιμετωπίσουμε με πρακτικό τρόπο και νομίζω ότι με μέτρα τεχνική συντήρηση και άλλα μπορούμε να βγάλουμε όλες τις απορρίψεις στην ε, στεριά. Και αν χρειαστεί να υπάρξουν και ε, αντισταθμίσεις, αυτό θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν σωστή προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά τις ε, μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Από ό,τι κατάλαβα, από σήμερα είναι υποχρεωτικό Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά ε, την επεξεργασία από το Συμβούλιο ε, ε, και, το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό θα σημάνει θανατική καταδίκη των μικρών παράκτιων περιοχών και των βιοτεχνιών εκεί και των ανθρώπων που ζουν από αυτή την δραστηριότητα. Εγώ έχω κάποια εμπειρία. Πραγματικά σας λέω θα σημάνει το τέλος αυτής της βιομηχανίας. Θα είναι χαριστική βολή οι μικροί παραγωγοί θα ε, εξαγοραστούν από μεγάλους παραγωγούς. Ε, λοιπόν, πρέπει να δούμε ε, πάρα πολύ προσεκτικά αυτό το θέμα των ποσοστώσεων. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στη χώρα σας, κύριε Πρεδρέφοντα, αλλά αν υπάρχει κοινή πολιτική, θα πρέπει η έλεγχη και οι κυρώσεις να είναι επίσης κοινέ. Αν έχουμε κοινό έλεγχο, δεν θα πρέπει να έχουμε και κοινέ κυρώσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές ε, παραβιάσεις, αλλά ε, μπορεί να γίνουν και εγκληματικέ ε, δράσεις. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα των κυρώσεων. Θέλω να ακούσω την άποψή της και για την κοινή δήλωση της δικής μου χώρας Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Βελγίου για το μελλοντικό χρηματοοικονομικό μέσο της κοινής πολιτικής για τη χρηματοδότηση του λευτικού στόλου. Είπε η Κομισιόν ότι δεν είναι υπέρ του να δαπανηθούν ε, άλλοι πόροι για τη χρηματοδότηση αυτού του κλάδου. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια ε, αποξήλωση, παροπλισμός ε, παραδείγματος χάρη. Εγώ θα μπορούσα να παροπλήσω το δικό μου ε, σκάφος, αλλά γιατί εγώ ή ένας άλλος να το κάνουμε αυτό, αν δεν έχουμε κάποια βοήθεια αν δεν μπορούμε να δώσουμε κίνητρα, να είναι πιο δελεαστική ο παραπλησμός κάποιων ε, σκαφών. Ε, νομίζω ότι κάτι ε, θα πρέπει να προβλέψουμε σχετικά. Τέλος. Αναφερθήκαμε και το πρωί σε αυτό και επανέρχεται τώρα. θα είσαι στα ενία αυτή την εποχή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε μέσα σε 6 μήνες ριζικά την πολιτική, αλλά εσείς νομίζω ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ε, στο θέμα των πόρων, του μερισμού των πόρων. Οι κοινοί πόροι, τα shared resources, σίγουρα ε, σε ό,τι αφορά τις παράκτιες χώρες, Νορβηγία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νύση, Φερόη, Ισλανδία, εκεί πρέπει να προστατεύσουμε και μπορούμε να προστατεύσουμε την αλία. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι μονομερώς ε, δρούν. Οπότε δεν πρόκειται να υπάρξει πλέον αλία και ο κύριος Στίβενσον το πρωί αναφέρθηκε στο Νταούκι uh, το Blue Whiting ναι, ναι, ναι. θα πρέπει κάποιος να αναλάβει ε, την ε, ιδιοκτησία αν θέλετε της όλης, ε, να αναλάβει τα ενία ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να δράσουν τάχιστα. Νομίζω ότι εκπροσωπώ τους περισσότερους όταν λέω ότι είναι απαραίτητη η συναπόφαση. Δεν μπορεί 900.000 ε, τόνοι να εκφορτώνονται, ενώ θα πρέπει να είναι 650.000 μόνο. Ε, διόρθωση της δερμηνέως Blue Whiting είναι το προσφυγάκι, όχι το νταούκι. Εγώ θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το σκουμπρί, δεν ξέρω ε, νομίζω ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα υπάρχει ένα σημαντικό ε, θέμα εκεί. Ε, οι αλλοί συμμορφώνονται πλήρως και έχουν δει και ωφέλη από αυτό και, τις στις τιμές το έχουν δει. Λοιπόν, με την αύξηση 150% είδαμε ότι η συνολική αξία παρακολούθησης θα χαμηλώσει και τις τιμές. Δεν θα αυξήσει κατά 150%. Λοιπόν, για το σκουμπρί. Eh, Θα σας δώσουμε 9,5 στα 10. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας την Πολωνική Προεδρία. Είναι η πρώτη φορά που η Πολωνία είναι Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Και μπαίνετε, αναλαμβάνετε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση. Όταν μεταρρυθμίζουμε την κοινή αγροτική πολιτική και τη γερική πολιτική. Εκπροσωπούσα τους πρασίνους, θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για το εξάμεινό σας. Όταν θα ηγείστε του Συμβουλίου και φροντίζοντας ότι αυτή τη φορά θα γίνει πράγματι η ριζική ε, μεταρρύθμιση που όλοι απαιτούν. Θα υπάρχει αντίσταση βέβαια από μελη από κάποια κράτη-μέλη. Θα συζητηθούν διάφορα θέματα. Σας εύχομαι καλή τύχη πραγματικά στις προσπάθειες να διαφυλάξετε τις προθέσεις μεταρρυθμίσεως περιβαλλοντική θέλουμε, κοινωνική και οικονομική βιώσιμη αληφτική πολιτική, τονίζοντας το περιβαλλοντική. Διότι αν δεν έχουμε αποθέματα και υγιείς ωκεανούς και επαρκή αποθέματα, δεν μπορεί να έχουμε οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη αλία και τομέα. Αδύνατον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυστηρότατοι. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη προοπτική στη διαχείριση των ε, αληφτικών αποθεμάτων. Διότι αν συνεχίσουμε με αιτήσιες προσεγγίσεις, τότε πάντα θα, δεχόμαστε τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη του ελευτικού τομέα και θα λησμονούμε τα μακροπρόθεσμα ωφέλη και για το περιβάλλον και για τον αληφτικό τομέα. Πρέπει να ακολουθούμε τις επιστημονικές συμβουλές. Είναι σημαντικότατο για μας. Ερώτημα. Τώρα έχει αποτελματωθεί η συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης στο Βυσκαϊκό Κόλπο. Έχουμε για ε, το γάδο κολλήσει. Τι θα κάνετε λοιπόν όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Διότι αυτά τα σχέδια είναι πολύ κρίσιμα για σωστή διαχείριση. Και αν δεν ξεπεράσουμε τα θεσμικά προβλήματα, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα να είναι βιώσιμη μεταρρύθμιση. Βιοπικιλότητα είναι το άλλο. Έχει φιλοδοξία η Πολωνική ε, Προεδρία τον Οκτώβριο να συμπεράσει το Συμβουλίο όσον αφορά τη στρατηγική για το 2020 για την βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον η θάλασσες και οι ωκεανοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι τουλάχιστον εξίσου μεγάλες εκτάσεις όσο και η χερσαία ε, έκταση και έχουμε 10 εκατομμύρια είδη στους ωκεανούς των, α, ε, της γης, περισσότερα από τα είδη τα χερσαία. Για να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα των ωκεανών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε. Είναι απαραίτητο. Αν το ξεχάσουμε στη στρατηγική θα ακολουθήσουμε, δεν είναι καν στρατηγική αυτή. Τι θα κάνει η Πολωνική Προεδρία λοιπόν, πώ θα ταιριάξει την διαμεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική με τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τη βιοπικιλότητα για το 2020. Χαίρομαι που τονίζετε ότι έχουμε διεθνή ε, υποχρέωση να συμμορφωθούμε με, τις διάφορες υποχρέωσεις που αναλάβαμε το 2015. Πρέπει να, να γίνει καταμέτρηση του πόσα ψάρια ε, μπορείς να βγάλεις από ένα συγκεκριμένο αλίευμα αλλά χρειάζεται και ηλικιακή δομή όσον αφορά τους ε, πληθυσμούς των ψαριών. Το λαμβάνετε υπόψη αυτό. Για τη μεταρρύθμιση της κοινής ελευθερικής πολιτικής και σε σχέση με τη βιοποικιλότητα. Μετά, εξωτερική πολιτική στην Αλία. Οι αλληλευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τι προτεραιότητες έχετε σαν Προεδρία και το Οικονομικό Ταμείο για την Αλία και τις επιδοτήσεις. Η Πολωνία και άλλες χώρες έχουν υπογράψει κοινή δήλωση ότι θα θέλετε να παραμείνει το ταμείο αυτό, το αλληλευτικό, το ευρωπαϊκό, στα ίδια επίπεδα όπως τώρα. Οι επιδοτήσεις, τι θα πρέπει να υποστηρίξουν κατά την άποψή σας. Οι πράσινοι πιστεύουμε ότι κάθε οικονομική στήριξη προς τον αληθικό τομέα είναι σημαντικό να οδηγεί σε μετατροπή, σε μετακίνηση προς πιο βιώσιμες ελευτικές πρακτικές. Να βοηθηθούν οι αλληλείς να μάθουν, να εκπαιδευτούν ή να βρουν άλλη δουλειά, εκείνοι που θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω της μεταρρύθμισης και της μείωσης του ελευτικού στόλου. κάθε οικονομική υποστήριξη θα πρέπει να ταιριάζει με τους στόχους κοινής ελευτικής πολιτικής, οικονομική, με τους οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς στόχους, κυρίως τους περιβαλλοντικούς. Είναι προαπαιτούμενο αυτό για τον ελευθερικό τομέα στο μέλλον. Αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις μου. Eh, για την e Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας κάνατε. Και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης. Η σημαντικότερη προτεραιότητα, ο σημαντικότερος στόχος φαίνεται να είναι μια μεταρρυθμισμένη και νέα ελευτική πολιτική που θα έχει αποτελέσματα για, τα, για τον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί θα επηρεάσει ε, τη βιωσιμότητα του κλάδου. Μιλήσατε για την περιφερειοποίηση. Όχι σήμερα, παλαιότερα. Σήμερα δεν επαναλάβατε αυτή τη λέξη. Δεν είπατε ότι είναι αναγκαίο να ε, γίνει περιφερειακή η διαχείριση των πόρων. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να το σημαντικότερο στοιχείο της εν λόγω μεταρρυθμισής. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Χωρίς περιφερειοποίηση, η μεταρρύθμιση αυτή δεν θα στεφθεί με επιτυχία. Οι απόπειρε μεταρρύθμισης, ε, ε, αποσπασματικά της κοινή αλληλευτικής πολιτικής όχι απλά δεν πέτυχαν τίποτα, το αντίθετο μάλιστα. Ουσιαστικά ε, κατέστρεψαν και τον ε, τομέα και τους πόρους και το περιβάλλον. Αυτές οι απόπειρες. Η Επίτροπος νομίζω ότι αυτό που θα μας πει σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να περιφεροποιούμε τώρα γιατί έχουμε τη σύνδεξη της αβώνας, ε, τις ε, νομοθετικές διαδικασίες, ε, θα βρει σίγουρα κάποιους λόγους για να μπλοκάρει τη διαδικασία περιφερειοποίησης. Και είμαι πεπισμένος ότι χωρίς αυτό το στοιχείο δεν πρόκειται να καταφέρουμε να αλλάξουμε την κοινωνιευτική πολιτική ούτε να δώσουμε στον κλάδο μια ευκαιρία να λειτουργήσει πιο πλασματικά και να μπορούμε να μεταλλευόμαστε ακόμη τους πόρους, τους αλληλευτικούς και να ζούμε από αυτούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το Σολομό και τα δίκτυα του Σολομού. Τα δίκτυα, συγγνώμη, του Σολομού. Έχει να κάνει με την ε, Βαλτική μόνο αυτό. Ή τίποτα με τη Βαλτική. Πιο πολύ με τη Μεσόγειο. Ουσιαστικά αφορά όλη την Ευρώπη. αλλιευτικά εργαλεία που οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ε, στη Μεσόγειο δεν επηρεάζει τη Βαλτική. Ο τρόπος αλήψης ε, του όλων. Πώς τελικά λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ότι δεν βλέπουμε ότι μπορεί οι αποφάσει που λαμβάνουμε να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις για μια συγκεκριμένη περιοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη μικρή παράκτη αλία, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για τον αλλιευτικό κλάδο που ζει σε καλή σχέση, συμβιωτικά με το περιβάλλον. Είναι οικογένειες που εργάζονται στη θάλασσα εδώ και πολλά χρόνια, ξέρουν να σέβονται τους αλλιευτικούς πόρους και νομίζω ότι θα έπρεπε την εμπειρία τους να την αξιοποιήσουμε γιατί η μικρή κλίμακα παράκτη αλία είναι και βάση τη πολωνική αλία. Έχουμε την εμπειρία στη χώρα μα. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε στην ε, παράκτη αυτή αλία να εξαφανιστεί. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι οι πιέσει ε, που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν. δεν ξέρω κι εγώ αν αυτές οι μεταφερόμενες, μεταβαζόμενες ποσοστώσεις ε, ε, θα φέρουν και το τέλος του ελληνικού τομέα. Ελπίζω να μην εισαχθούν στην κοινή ελληνική πολιτική. Και σε ό,τι αφορά τέλος της απορρίψης, είναι το όνειδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από κάποια προγράμματα τα οποία μετέδωσε η Βρετανική τηλεόραση BBC, νομίζω ότι ε, έχει γίνει αντιληπτό τι εστί απόρριψη, τι εστί απορρίψεις και υπάρχει πραγματικά ε, ντροπή για αυτό το φαινόμενο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, στη Βαλτική ε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μπορούν ε, τα πλατέα ψάρια στη Βαλτική να απορρίπτονται γιατί μπορούν να επιβιώσουν στο νερό, αλλά σε ό,τι αφορά τον ε, βακαλάο, το γάδο, νομίζω ότι πραγματικά είναι έγκλημα η απόρριψή του. Είναι πολύτιμο ε, είδος, δυστυχώς δεν μπορεί να επιβιώσει όμως με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, βιομηχανική αλία. Αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στη Βαλτική, αυτή η δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, έχει τη μεγαλύτερη ποσόστοση στην αγορά της Βαλτικής. Αλλά ταυτόχρονα καταστρέφει το περισσότερο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το περιβάλλον σε θάλασσα αυτή. Έχω και τα στοιχεία μιας ανάλυση στη διάθεσή μου. Ότι η βιομηχανική αλληλεία στη Βαλτική εξαλείφει ουσιαστικά τους αλληλευτικούς πόρους, ιδίως στη Δυτική Βαλτική. Η Ρέγκα μάλλον ο γάδος σχεδόν έχει εξαφανιστεί και αυτό πολλοί λένε ότι οφείλεται στη βιομηχανική αλία. Και επίσης έχουμε και προβλήματα πολύ σημαντικά με τη ρέγγα που στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκή Ένωσης δεν θεωρούνται, ε, δεν καταναλώνονται πάρα πολύ. Εξαφανίζονται επίσης ε, πολλά ψάρια τα οποία χρησιμοποιούνται και ως δόλωμα κυρίως ή ως ε, ηχθιάλευρα. Πρόκειται για κάποια ψάρια τα οποία είναι πεντανόστιμα αλλά τα χρησιμοποιούν πολύ ως ηχθιάλευρο. Τα πελαγικά είδη όμω, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο για την ε, κατανάλωση από, ε, από τον άνθρωπο. Ε. Λοιπόν, κοιτάξτε, λέει η πρόεδρο, δεν είναι, επαναλαμβάνω εδώ ο υπουργό που την ιδιότητά του ω Πολωνού Προέδρου, αλλά ω προέδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο. Ξεκινήσαμε ήδη από τις 8.30 με τους συντονιστές. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι πέντε συνάδελφοι που θέλουν το λόγο και θα τους παρακαλέσω να μην κάνουν ε, ομιλίες, αλλά ερωτήσεις. Και να πω επίσης, πρέπει να είμαστε σύντομοι, γιατί πρέπει ε, να φύγουμε σε κανένα δεκάλεπτο με τον ε, Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω πολύ χρόνο. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα των ερωτήσεων που έχουν σχέση με τη Βαλτική. Ιδιαίτερα για τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης του γάδου. Ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Η κατάσταση των αποθεμάτων μάλιστα είναι τόσο καλή που αποτελεί κίνδυνο για τα αποθέματα σαρδελόρεγκας. Ξέρουμε ποια είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ειδών, γάδου και σαρδελόρεγκα, και έχει νόημα όταν αυξάνεται τόσο πολύ ο πληθυσμό γάδου να έχει αρνητικέ επιπτώσει. στον πληθυσμό της ε, σαρδελόρεγκα. Ακούσαμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μια λύση Διαφορετικά καταστρέφεται η διατροφική αλυσίδα και θα έχουμε τεράστια προβλήματα λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο ειδών. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τη γνώμη του κυρίου Υπουργού σχετικά με την αύξηση κατά 40% των αποθεμάτων γάδου. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης του γάδου υπάρχει έχει καθοριστεί και η αλληλευτική ικανότητα και νομίζω ότι με τα κατάλληλα επιστημονικά δεδομένα μπορούμε να καταλήξουμε στα εθνικά στοιχεία που πιστεύω ότι πρέπει να είναι αύξηση της αλληλευτικής ικανότητας για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ. Ραούλ Ρωμέβα, μας πρέπει να Πρόεδρος. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Τονίσατε την ε, υδατοκαλλιέργεια, την ηχθειοκαλλιέργεια. Αλλά δεν μας ε, δώσατε περισσότερες διευκρινήσεις. Μιλάτε για τη βιωσιμότητα των πόρων, γιατί τότε δεν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή και γιατί ε, πόροι μεταφέρονται σε μια άλλη δραστηριότητα ενώ θα ήταν καλύτερο να ε, βασιστούμε στην ε, διατήρηση των πόρων στο φυσικό τους περιβάλλον και δεύτερον πολλά ψάρια, μεγάλη ποσότητα που αυτό τελικά είναι και επιβλαβές για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Και ένα δεύτερο ερώτημα σε ό,τι αφορά τον επαναπροσδιορισμό του κλάδου θα με ενδιέφερε Μάλλον με ικανοποιεί βλέποντας ότι οι στόχοι του Johannesburg ε, του 2015 δηλαδή είναι στην ε, ημερήσια διάταξη και αυτός είναι ένας σαφής στόχος. Αυτό βέβαια συνεπάγεται τις θυσίες ε, του κλάδου. Δεν μπορεί να γίνουν έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προβείτε σε αυτή την διάταξη και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβουμε για τον επαναπροσδιορισμό του κλάδου, για να δούμε ποιος θα έχει ε, δικαίωμα ε, να αλλιεύει και ποιος θα εξαιρείται αυτού του δικαιώματος. Ευχαριστούμε ο κύριος Στίβενσον. Κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε... Προεδρεύοντα, τα τελευταία δύο χρόνια επανειλημμένα ακούσαμε την Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, να λέει ότι η κοινή πολιτική υπό την μπορούσα μορφή τη ήταν μια καταστροφή. Το ακούσατε αυτό από πολλούς από τους σημερινούς αγορητές. Μας είπε επίσης επανειλημμένα ότι πολεμούσε κατά των ίδιων νομικών της συμβούλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είπαν ότι το στοιχείο της περιφερειοποίησης που ζητήσαμε στο Κοινοβούλιο για όλες, όλες οι πολιτικές ομάδες ζητήσαμε αυτό, όταν συζητήσαμε την Πράσινη Βίβλο, ότι αυτό το στοιχείο της περιφερειοποίησης θα εστρέφεται κατά της συνθήκης. Άκουσα φήμες και πολλοί από εμά ακούσαμε παρόμοιε φήμες, σύμφωνα με τι οποίε η περιφερειοποίηση στο πακέτο τη έχει αποδυναμωθεί, δηλαδή οι γραφειοκράτε νίκησαν με άλλα λόγια. Αν περί αυτού πράγματι πρόκειται, Υπουργέ, βασιζόμαστε σε εσά και στη συνεργασία σας μαζί μας που υποσχεθήκατε το πρωί, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε το ότι το στοιχείο της περιφερειοποίησης θα αποκατασταθεί πλήρως. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την καταστροφική μικροδιαχείριση από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Σκασίλα μου να αναφέρεται αυτό συνθήκη ή όχι. Κατέστρεψε την αληφτική συμφωνία, κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και δεν θα δεχθούμε τίποτα λιγότερο από ότι μια περιφερειοποίηση η οποία θα έχει νόημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα, δεν θα μιλήσω επί μακρόν, διότι χθε μπόρεσα να μιλήσω και να συγχαρώ τον Υπουργό κατά τη διάρκεια μάλλον του πρωινού της Επιτροπής Γεωργίας. Έχω το εξή ερώτημα λοιπόν. Ε, έριξα μια ματιά στο έγγραφο της Προεδρίας που αναφέρεται στις προτεραιότητες σας. Χρονολογείται 1η Ιουνίου αυτό το έγγραφο. Λέτε ότι η εξωτερική πολιτική για την, κοινή, για την αλληλευτική πολιτική, για τον τομέα έχει ως εξής οι στόλοι μακράς αποστάσεως λειτουργούν σε διαφορετικό πλαίσιο και είπατε ότι χρειάζεται να απελευθερωθεί η διαχείριση αυτού του τομέα. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό που αναφέρει το έγγραφο. Τι σημαίνει αυτό που διάβασα, σημαίνει αυτή η φράση απελευθέρωση της διαχείρισης των ελευτικών στόλων μεγάλης απόστασης. Ε, Σας ευχαριστώ. Η κυρία που ήταν να πάρει το λόγο δεν είναι εδώ. Λοιπόν, θα σας δώσω, κύριε Υπουργέ, τότε αμέσως το λόγο να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι να δίνω το να μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις ε, σε τόσο λίγο χρόνο. Ας πω ότι μπορώ πάντως. Νομίζω ότι περισσότερο από εσά ε, κάνατε ρητορικέ ερωτήσει, δηλαδή δώσατε και την ερώτηση και την απάντηση ταυτόχρονα. Σίγουρα πάντως είναι σημαντική η συζήτηση γιατί μας προετοιμάζει στη μεγάλη αυτή ε, μεταρρύθμιση. Έχουμε την ίδια Κομισιόν, το ίδιο Συμβούλιο, αλλά ε, δεν βλέπουμε την ίδια συμπεριφορά. Εμένα μου αρέσει η στάση του Κοινοβουλίου. Η μεταρρύθμιση του 2002 απέτυχε. Κατέστρεψε τις αληφτικές δυνατότητες, κατέστρεψε τον κλάδο και τους φυσικούς πόρους ταυτόχρονα. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι αυτή η νέα μεταρρύθμιση πρέπει να είναι πιο βαθιά. και στην κοινή γεωργική πολιτική γίνεται λόγο για μεταρρύθμιση, για ανάγκη μεταρρύθμιση. Ακούμε και εκεί κάποιε φωνές που λένε ότι θα πρέπει να είναι πολύ απότομη μεταρρύθμιση, ότι ούτε η Αλία ούτε η Γεωργία μπορούν να, να αντέξουν μια επανάσταση. Εγώ ακούω τις απόψεις σας. Πρέπει να γίνουν αποφασιστικές αλλαγές. Θέλω να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να τεθεί πλήρως σε ισχύ. Μιλώ για τη διαδικασία της συναπόφασης. Η ανταλλαγή απόψεων κατά την επόμενη εγγράφων πρέπει να είναι πραγματική ανταλλαγή. Ο κύριος Στίβενσον είπε ότι από τη μία μας λένε ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε περιφερειοποίηση, ε, αυτό ε, δυνάμει της συνθήκης, και από την άλλη ακούμε ότι οι γραφειοκράτες δεν την ε, περιλαμβάνουν αυτή την ιδέα της περιφερειοποίησης στα δικά τους τα έγγραφα. Δεν μπορώ να προτρέξω, θα ήθελα να ακούσω και τι θα πει η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη. Βέβαια, σίγουρα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μόνο των πολιτικών και των γραφειοκρατών, οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί. Εμεί πρέπει να κάνουμε το βήμα προ τα εμπρό. Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των πόρων και μάλιστα την ορθολογική διατήρηση των πόρων, Ναι, λέγεται ότι δεν είναι 100% αξιόπιστες οι επιστημονικές ε, αναλύσεις. Αυτό αληθεύει. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες ούτε και σε ό,τι αφορά τα πραγματικά λιεύματα. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αδήλωτης παράνομης άναρχης αλίας. Μεταρρύθμιση του 2002 δεν στέφθηκε με επιτυχία γιατί δεν την αποδέχθηκε ο κλάδος. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά εμείς οι πολιτικοί πρέπει να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον κλάδο. Να συζητήσουμε δηλαδή με τους άλλους, να τους ε, εξηγήσουμε τα πράγματα. Γιατί αν αυτοί δεν αποδεχθούν αυτή τη μεταρρύθμιση, τότε για μια ακόμη φορά θα αποτύχει. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν δεν είναι μόνο το μαστίγιο. Χρειαζόμαστε και το καρότο. Και αυτή τη φορά το καρότο θα είναι η ενημέρωση, η συζήτηση. Και κάτι ακόμη. Στους έξι αυτούς μήνες εγώ έχω το ρόλο του συντονιστή. Φυσικά και έχω τις δικές μου εμπειρίες και τις δικές μου απόψεις. ούτε καν με ενδιαφέρει το ότι ασκώ την Προεδρία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Απλά με την ιδιότητά μου αυτή, εγώ θα πρέπει να βρω ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιφερειοποίηση. Ναι, πράγματι πρέπει να της δώσουμε μια ευκαιρία. και σίγουρα πρέπει να μας απασχολήσει η βιομηχανική αλία. Πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Γιατί πράγματι δεν ε, είναι ευεργετική ούτε για τον ε, αλία ούτε για τον ανθρώπινο παράγοντα στην αλία γενικά. Και σε ό,τι αφορά την ορθολογική διαχείριση, έχουμε το πρόβλημα της υπεραλίευσης σε άλλα μέρη του κόσμου και πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να εκπονήσουμε κάποιο μηχανισμό, κάποιο σύστημα ε, αμοιβαίου ελέγχου με τους ε, εταίρους μας, όπως είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, τα νησιά Φερόε ή και η Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα Έχουμε δύο κράτη-μέλη που πρέπει να δεχθούν τους κανόνες της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Τα υπόλοιπα παρακτία κράτη όμως, τα οποία ε, διαβρέχονται από την ε, Μαύρη Θάλασσα, δεν δίνουν δεκάρα, για να το πω έτσι, για όλες αυτές ε, τις προδιαγραφές και για όλους αυτούς τους κανόνες. Άρα πρέπει και να θεσπίζουμε πρότυπα και κανόνες, αλλά ταυτόχρονα να φροντίσουμε να μπορούν να εφαρμόζονται. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εμά, αλλά ισχύει και για του εταίρου μα από τρίτε χώρε. Ω Προεδρεύον του Συμβουλίου, θέλω, όπω είπα, να έχω το ρόλο του συντονιστή. Δηλαδή πρέπει να ακούω τι μου λέτε εσείς, γιατί πιστεύω ότι εσείς είστε πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα του κλάδου. Σίγουρα πολύ κοντύτερα από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. από τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πετύχουμε ως Προεδρία. Είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει για το 2015, αλλά αυτό να το κάνουμε με ηρεμία, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχείρηματα όλων των πλευρών. Πάλι να, την, να αναφερθώ στην περιφερειοποίηση. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεις ε, της Μεσογείου, της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας, για συγκεκριμένα ήδη μίλησαν κάποιοι από εσά. Πράγματι, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι η επίλυση των ζητημάτων αυτών να γίνει περιφερειακά, σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, προς τούτο πρέπει να είμαστε να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί ο τομέας και ο κλάδος σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ε, τι θα πλήξει περισσότερο, ποιοι θα φυγούν από τις αποφάσεις μας, πιο πολλοί παρά οι εφοπλιστές ή οι πλειοκτήτες. Εγώ θέλω να έχουμε μια συζήτηση όλοι μαζί εδώ και να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερη. Όταν λοιπόν μίλησα για την εκθεοκραλιέργεια, αναφερόμουν και για την εκτοκαλλιέργεια στη θάλασσα αλλά και στην υπηρετική χώρα την οποία δεν προσέχουμε ιδιαίτερα. Θέλουμε να εξοικονομήσουμε, θέλουμε να προστατεύσουμε τους θαλάσσιους πόρους, ε, τους πόρους, ε, τους ε, των ωκεανών. Αλλά σίγουρα στην υδατοκαλλιέργεια, στην δεν θα πρέπει να ε, αφιερώσουμε να αποδώσουμε όλους τους πόρους, όλα τα κονδύλια. Εδώ πάντως πρέπει να ολοκληρώσω την σημερινή μου παρέμβαση. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τι ερωτήσει και για τη συζήτηση που είχαμε και να σα πω ότι πρέπει και, γίνεται σεβαστή πλήρωση στην απόφαση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σα ευχόμαστε καλή τύχη. Πρέπει να φύγουμε εμείς και θα παρακαλέσω τον κύριο Στίβενσον να με αντικαταστήσει, εάν έχει την ευγενή καλοσύνη. Okay, ladies and gentlemen, uh, the chairman... Λοιπόν, κύριε και κύριοι, έπρεπε να, πάει, να φύγει για συνέντευξη τύπου η Πρόεδρος μαζί με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Οπότε, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. If we could move on with item... Να προχωρήσουμε και πάμε στο σημείο 12 της ημερήσιας ε, διάταξης σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσια που υπογράφθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διευθυντής που καθορίστηκε από την Υπηρεσία Ελέγχου της Αλληλείας του Βίγκο πρέπει να εμφανιστεί στην Επιτροπή μας για την απόψεων όσον αφορά τις δραστηριότητε και πρόγραμμα εργασιών της υπηρεσίας. Με τα χαράς βλέπουμε σήμερα το πρωί ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο, τον υποψήφιο διευθυντή, τον κύριο Πάσκαλ Σαβαρέ, μάλλον τον προσφάτως οριστέτα διευθυντή. Λοιπόν, ευχαριστώ τον προκάτοχο του κ. Σαβαρέ, τον κύριο Κώστερ, που υπηρέτησε ως διευθυντής της υπηρεσίας. Τον ευχαριστούμε για τη σκληρή δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Βεβαίως δημιούργησε την υπηρεσία από την αρχή, από το μηδέν, θα θυμόσαστε ότι μέλη της Επιτροπής Αλίας πήγανε στο Βίγκο σε αντιπροσωπεία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον κύριο Κώστερ στο Βίγκο στην Υπηρεσία Ελέγχου της Κτιμούμε εκτιμούμε τις προσπάθειες που κατέβαλε και φεύγει από, έχοντας αφήσει αυτή την υπηρεσία ελέγχου της Αλίας σε πλήρη λειτουργία και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε καλές σχέσεις με τον κύριο Σαβαρέ όπως είχαμε καλές σχέσεις με τον κύριο Κώστα. Παρευθείς, δίνω το λόγο με τα χαράς στον κύριο Σαβαρέ για να μας μιλήσει. Για να μας ενημερώσει επί των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας ελέγχου της αλίας του Βίγκο. Έχετε το λόγο κύριε Σαβαρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Είναι χαρά. Και θα ήθελα να σας μιλήσω. Ανήκω στη γαλλική διοίκηση. Πρώην ναυτικός ταξιωματικού. 15 χρόνια ήμουν στη θέση πριν μπω σε διοίκηση. Έχω εμπειρία από επιχειρήσεις θαλάσσιες. Ήμουν ειδικό στα ραντάρ και ηλεκτρονικό πόλεμο. Ειδικό για τον έλεγχο ναρκών μετά ήμουν διοικητής ενός κέντρου διάσωσης, θαλασσίας διάσωσης και επίσης ε, σε μια υπηρεσία διαχείρισης ε, κίνησης θαλάσσιας. Ήμουν επί 26 χρόνια στη γαλλική διοίκηση. Ασχολιόμουν με έλεγχο και επιθεωρήσεις. Με ενδιαφέρει πολύ διαχείριση μιας υπηρεσίας Καθήκον μου είναι να είμαι διαφανής απέναντί σας, διότι εκπροσωπείτε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και έχω καθήκον απέναντί σας και απέναντι στο λαό που εκπροσωπείτε. Να είμαι σαφής πρέπει, να είμαι διαφανής και να σας δίνω τις καλύτερες πληροφορίες όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθεί η υπηρεσία μας. Το βιογραφικό μου ε, είμαι από τη Βρετάνη, από τη Γαλλία, από μικρή κοινότητα. Όταν γεννήθηκα η Αλία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Νησί στην νότια ακτή του Γιούρα. Και ξέρω τα βρετονικά και τα γαλλικά. Έχει πολύ ισχυρή ταυτότητα αυτή η περιοχή της ε, Ευρώπης. όσον αφορά την υπηρεσία. Είναι πολύ αποδοτική. Διότι όπως είπε ο Πρόεδρος, το σύστημά μας είναι πολύ αποτελεσματικό. Το ξεκίνησε ο κύριος Κώστερ. Δημιούργησε την υπηρεσία από το μηδέν. Μπόρεσε να αναπτύξει ένα πολύ καλό σύστημα βάση της διαχείρισης των κοινών αληφτικών επιχειρήσεων και σχετικών σχεδίων κοινού ελέγχου. Πιστεύω προσωπικά, άμα επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτό επί μερικά λεπτά, θα ήταν να τονίσω το ότι θέλουμε να έχουμε κώδικες συμμόρφωσης για τα κάτι μέλη, ώστε να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας πολύ καλά την οικονομική κατάσταση γνωρίζοντας ότι χρειάζεται να γίνουν μεγάλες οικονομίες όσον αφορά τα χρήματα της κοινότητας και των κρατών μελών. Χρειάζεται συντονισμός επιχειρήσεων. Με αυτό σχολείται η υπηρεσία. Τρεις στόχους έχουμε. Σαφής ελέγχους, δείκτες, βαθμολόγηση, στόχους όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας, δημιουργία δυναμικού και βοήθεια των κρατών μελών. Καθήκον μου είναι πολύ αποδοτική σχέση με τα κράτη-μέλη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις τους και τις ανάγκες τους. Θέλουμε να είμαστε στο δυνατόν πιο αποδοτικοί με τα χρήματα τα οποία θα μας δώσετε. Διότι είστε ο ισχυρότερος κλάδος της δημοσιονομικής αρχής, της αρχής του προπολογισμού. Όσον αφορά τη βοήθεια των κρατών μελών, η κατάσταση εκεί είναι πολύ διαφορετική. Κάποια κράτη-μέλη χρειάζονται βοήθεια για τη βελτίωση της κατάρτισης για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων, τη διασταύρωση στοιχείων. Χρειάζονται σωστές τεχνικές, χρειάζεται απόδοση όσον αφορά του έλεγχους και τι επιθεωρήσεις στον τομέα τη αλληλεία. Όσον αφορά την παράνομη αλληλεία. είναι κατάρα για όλους, μάστιγα, για τη βιομηχανία και για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Περιμένει πολλά από μας ο λαός. Τι κάνουμε για την καταπολέμηση του προβλήματος. Θα είμαστε αναποδοτικότεροι στην καταπολέμηση της παρανομαλίας με νέα εργαλεία που θα διασταυρώνουν στοιχεία ας πούμε στοιχεία Frontex, ε, Interpol, διότι συνήθως ε, η παράνομη αλία πραγματοποιείται από το διεθνές ε, έγκλημα. Αυτά για να βρούμε μια σωστή απάντηση. Ε, και αυτά για να μην μακρηγορήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σάβαρε. Ελπίζω στο ρόλο αυτό να έχετε αποτελέσματα και να περάσετε όμορφα. Ένα μέλος της Επιτροπής θα να πάρει το λόγο. Η κυρία Λαβέ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Σάβαρη. Έχετε πολύ σημαντικό καθήκον μπροστά σας στην υπηρεσία ελέγχου της Αλίας και μιλώ εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής Αλίας του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η υπηρεσία για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειες τους όσον αφορά τους ελέγχους και όπως είπε ο κύριος Στίβενσον επισκεφθήκαμε το Βίγκο πέρσι εντυπωσιαστήκαμε από αυτά που είδαμε όσον αφορά τα κοινία σχέδια δράσης στη Βαλτική και στη Μεσόγειο για τον τόνο υποστηρίζουμε τις αστηριότητες της υπηρεσίας Είμαι εισηγήτρια για μια έκθεση το πώς θα μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση παρανόμου αλληλείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι η ευθύνη της Ένωσης δεν είναι μόνο να καταργηθεί, να σταματήσει η παράνομη αλληλεία εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά εφόσον είναι μεγάλος παράγων στην αλία Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλα μέρη του κόσμου, και εισάγουμε πολλά μεγάλες ποσότητες στην Ένωση, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σαν ένα από τα πιο πλούσια μέρη του κόσμου, πρέπει να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παρανομαλίας στον κόσμο. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας. Πώς λοιπόν η υπηρεσία σας μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. η υπηρεσία σας πώς να το πω θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο ελέγχοντας τα ύδατα εκείνα στα οποία, τα οποία καλύπτονται από ληφτικές συμφωνίες. Έχουμε κοινοτικά μισθωμένα σκάφη, κοινοτικό μισθωμένο σκάφος που κάνει και ερεύνες σε διεθνή ύδατα. Μπορεί αυτό κατά την άποψή σας να ε, μεγαλώσει τα δραστηριότητα, να επεκταθεί. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει σε διεθνές επίπεδο την παράνομη αλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Λαβέν, και άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Κουν είναι ο πρώτος από τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαβαρή. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία η υπηρεσία σας ε, κινείται γίνονται προσπάθειες όχι μόνο στην καταπολέμηση της ε, αλληλείας της παρανόμου αλλά και έχει άλλο ένα σημαντικό καθήκον που είναι ο συντονισμός των αλληλευτικών αρχών των κρατών μελών. Και συζητούμε την κοινή αλληλευτική πολιτική για την επόμενη επταετία και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σαν μέλη του Κοινοβουλίου και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικρινόμεθα από τους ε, αλληλείς διότι υπάρχει ένα ολόκληρο ελεγκτικό δίκτυο ε, με ηλεκτρονικά μέσα, με στοιχεία που συλλέγονται και από τηλέφωνα, ε, συλλογή πληροφωνίων που επεκτείνεται σε όλο τον τομέα κάθε σκάφος έχει άδεια. Χρειάζεται άδεια για να βγει στην ανοιχτή θάλασσα το σκάφος. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Και το σημείο είναι συγκεκριμένο που γίνονται εκφορτώ στα κράτη-μέλη. Και οι υποπτικές αρχές είναι υπεύθυνε και γι' αυτό. Μετά έχουμε και ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου που στο μέλλον θα συμπεριλαμβάνει τα τάκ για κάθε σκάφος. Το μπλε τετράγωνο, το μπλε κουτί θα γίνει και αυτό ηλεκτρονικό. Το ξέρετε, είστε ειδικό όσον αφορά τα ναυτικά θέματα, είχατε σχέσεις πολλές με τα ηλεκτρονικά και στην ε, Γερμανία και τηλεφωνάει ο κόσμος στα αρχές και τους λέει που είναι. Τηλεφωνούν οι ψαράδες αν χρειάζονται το ηλεκτρονικό ε, πλοίου ή όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Χρειάζεται να υπάρχει μια καλή βάση για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θεσπίζονται και εφαρμόζονται. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν οι αλλοί σε λάθος περιοχές. Θα πρέπει να είναι λογικά τα τάκ. Θα πρέπει να προστατεύουμε τις θάλασσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα εξετάσει αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Θα πρέπει να καταλήξετε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, ούτω ώστε η αλληλευτικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποπτεύεται σωστά όσον αφορά το μάτι των δικτυών, παραδείγματος χάρη, με τα ΤΑΚ, και εποπτεία και έλεγχος τρίτων χωρών είναι κάτι που επίσης ε, απαιτείται τι κάνουν οι Ισλανδοί, τι γίνεται στις νήσους Φερόες, τι γίνεται με τη Ρωσία στη Βαλτική και στον Ατλαντικό και με την Νορβηγία. Όλα αυτά είναι παραδείγματα, έτσι δεν είναι, είναι πάντα παραδείγματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ανακαλύψω τι δυνατότητες υπάρχουν για τους ελέγχους, ε, αν είναι θέμα ποσοστώσεων ή όχι. Πρέπει να εστιαστούμε πραγματικά επί ενός σαφού συστήματος, ξεκάθαρου συστήματος εντός των κρατών μελών, αλλά επίση θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα ελέγχου σαφέ για τον έλεγχο τρίτων χώρων. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Ο κύριο Γκαμπάτσεκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σα καλωσορίζουμε και σα συγχαίρουμε για την ανάληψη των πολύ σημαντικών καθηκόντων σα. Όπω είπε ο κύριο Κούν, η υπηρεσία ελέγχου είναι εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής αλληλείας. Θα μπορούσα να παραθέσω πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τη δραστηριότητα των αρχών μέχρι τώρα και θα θέλαμε ε, να μιλήσουμε και για τις απόψεις μας σχετικά με το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ο οργανισμός στο μέλλον. Σημαντικό είναι η ανάληψη της ευθύνης. Θα πρέπει 100% να αναλάβει την ευθύνη η υπηρεσία ελέγχου σχετικά με τις ε, δραστηριότητες της αλίας. Είμαι πεπισμένο ότι υπό την ηγεσία σας η κοινοτική υπηρεσία ελέγχου θα λειτουργήσει σωστά και αυτό οφείλεται και στο ιστορικό σας, γιατί το βιογραφικό σας και αυτά τα οποία μας είπατε μας έχουν πείσει ότι έχετε την εμπειρία, ήσασταν υπεύθυνο για τη διάσωση ανθρώπινων ζώων και τώρα θα είστε υπεύθυνο για την διάσωση του μέλλοντος της αλίας. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Σας παρακαλώ να ε, μην ε, ε, ενδώσετε σε πολιτικές πιέσεις, να αντιμετωπίσετε όλες τις χώρες με βάση την αρχή της ισότητας, γιατί πραγματικά αυτό χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε μια κοινοτική πολιτική αλληλείας, χωρίς να δίνουμε λιγότερη ή περισσότερη σημασία σε διάφορες χώρες. Άλλη μια σημαντική αρχή είναι η αρχή της διαφάνειας οι πληροφορίες ε, που φτάνουν στην υπηρεσία ελέγχου νομίζω ότι είναι πληροφορίες που μπορούν να δίδονται και στην κοινή γνώμη και οπωσδήποτε πρέπει να δίδονται σε εμά του ευρωβουλευτέ. Είμαι βεβαισμένο ότι θα λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπηρεσία ελέγχου. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκραμπάτσεκ. Η κυρία Άντρε Μπαρία έχει το λόγο τώρα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για τον ορισμό σας στην κεφαλή μιας πάρα πολύ σημαντικής υπηρεσίας και χαίρομαι γιατί θα μείνετε στο Βίγκο. Ε. Πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Είναι και πάρα πολύ όμορφη πόλη και θα φάτε πολύ καλά εκεί. Καλό είναι να κάνει κανείς διαφήμιση στην Ισπανία. Αναφερθήκατε στη συνεργασία των κρατών μελών. Αυτό για μένα είναι ζωτική σημασία. Μιλήσατε για την ενημέρωση, για την ποιότητα των δεδομένων. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται απόφαση να γίνεται ανάλυση χωρί ποιοτικά δεδομένα. Χωρί επίση ομοιόμορφα ε, ε, δεδομένα τα οποία αξιολογεί κανεί με τον ίδιο τρόπο και αν δεν υπάρχει και κάποια προβολή. Η υπηρεσία του Βίγκο αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει είναι να επιβάλλει κυρώσει αν δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ κράτων μελών. Ποια, πώς θα φροντίσετε να γίνονται σεβαστέ οι κοινοτικοί κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο απαιτητικό θέμα. Υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία που έχουν ε, αδύνατα σημεία σε ό,τι αφορά ε, την ε, πανομοιαλία και κάποιες φορές έχουν ε, μία φήμη που άλλοτε είναι δικαιολογημένοι, άλλοτε όμως όχι. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς πώς μπορείτε εσείς να επιβάλλετε στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ε, τα πρότυπα ελέγχου, τους κανόνες ελέγχου που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Άντες Παρέα. Να προσθέσω κι εγώ κάνα δύο πράγματα κύριε Σαβαρέ. Όταν επισκεφτήκαμε το Βίγκο ενδιαφερθήκαμε βλέποντας ότι συγκεντρωνόταν στον ε, τόνο τον, ε, η όλη προσπάθεια. Σύντομα μετά την επίσκεψη όμως η κρίση από την υπερεκμετάλλευση του βορειοατλαντικού ε, Ατλαντικού όσον αφορά τον Μπακαλιάρο, το Άδα αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε. Το έθεσε ο κ. Κούν το πρωί αναφέρθηκε στην Ισλανδία και στην ίσως Φερόες που αυθαίρετα αύξησαν το αλλιευμά τους στις 150.000 τόνους ο καθένας. Περίπου ένα εκατομμύριο τόνοι θα, σκουμπριού θα αλλιευτούν φέτος και θα υπονομευθεί ε, το απόθεμα. Δεν θα μπορεί να επιβιώσει το σκουμπρί. Δεν θα είναι βιώσιμο απόθεμα αν συνεχιστεί αυτή η αλληλεία, η αλίευση. Δυστυχώς τα επιχειρήματά μας όσον αφορά το τι κάναμε εμείς για την προστασία του αποθέματος σκουμπριού στην Ευρώπη υπονομεύθηκε η πολιτική μας αυτή διότι ο στόλος της, του κράτους μέρους του δικού μας της Σκοτίας συνελήφθη να κάνει παράνομες εκφορτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σκουμπριού. Και πιο πρόσφατα ο Ισπανικός στόλος βρέθηκε ένοχος τέτοιας παράνομης εκφόρτωσης της τάξης περίπου 100.000 τόνων ε, σκουμπριού. Ε, οπότε εμείς τώρα τι να πούμε ότι εμείς διαφυλάσσουμε τα αποθέματα του σκουμπριού όταν τα κάναμε αυτά. Στείλαμε μια κοινή επιστολή κάποια μέλη της Επιτροπής. Υπογράψαμε λοιπόν μια επιστολή και τη στείλαμε στην υπηρεσία του Βίγκο, στον κύριο Κώστα και ζητήσαμε να αναλάβει δράση η υπηρεσία. Και τι μας είπαν, ότι ο εσωτερικός κανονισμός απαιτούσε έτοιμα, αίτηση κράτους μέλους με την υποστήριξη του Συμβουλίου των Υποργών. Και ήταν μια έκπληξη ότι ο εσωτερικός κανονισμός είναι αρκετά άκαμπτος. Ε, δηλαδή, αν διαπιστώσεις ότι υπάρχει παράνομη δραστηριότητα ακόμα και στα είδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορείς να κινηθείς ε, χωρίς συγκεκριμένη άδεια ε, του Συμβουλίου. Μπορείτε να επεκταθείτε από αυτού. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνατε για το θέμα του, σκουμπριού. Ε, και λόγω δραστηριότητα Ισλανδίας και νήσων θερών και τα οκτώ αποθέματα του σκουμπριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούνται βιώσιμο αλίευμα είναι πιστοποιημένα ότι πρέπει να ακολουθείτε, ε, είναι αλίευμα το οποίο πρέπει να ακολουθείτε συγκεκριμένη ε, ε, απόδοση αλληλευτική. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να ελέγξουν οι αλληλείς μας όσον αφορά το πρόβλημα. Και αυτό είναι τραγικό. Χρειάζεται να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνουν κάτι δική μας αλληλείς για αυτά που κάνουν οι Ισλανδοί και οι νήσοι Φερόες. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι κάτι θα γίνει ούτως όσο σταματήσει η παράνομη αλληλεία του σκουμπριού στα νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μπορείτε να κάνετε κάτι ε, ούτω ώστε να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργούν η Ισλανδία και οι νήσοι Φερόες. Βέβαια δύσκολο αυτό. Ε, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες διαβεβαιώσεις πάνω σε αυτά. Πολλά έχετε, πολλές ερωτήσεις έχετε να απαντήσετε και σας δίνω το λόγο. Euh, Monsieur le Président. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσω να μιλήσω και ισπανικά προς την κυρία Ανδρέας Μπαρέα. Όσον αφορά τις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δυνατότητα ε, εποπτείας και ελέγχου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία, ιδίω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η αξιοσημείωτη δουλειά την οποία έχει ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οποία έχει επικυρώσει το Συμβούλιο για τον κανονισμό 2005 του 2008 που θέσπισε κανόνες και υποχρεώσεις ε, για ε, την ανιχνευσιμότητα ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο κατά της παράνομης και άναρχης αλίας. Νομίζω ότι δεν έχουμε ακόμη επιτύχει τους στόχους μας σε σχέση με το εργαλείο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δουλεύει μαζί με τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να διαμορφώσει καλύτερα αυτό το εργαλείο. Και ε, αν δούμε τι κάνουν άλλα κράτη όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς στο πλαίσιο ε, του δικτύου MCS, και με τον έλεγχο του κράτους λιμένα νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελεσματικά μέτρα και μπορούμε να συνεισφέρουμε στην μείωση των παράνομων αλλιευμάτων. Δεύτερον, όπως είπα προηγουμένως, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία με τα αντίστοιχα μέτρα, δηλαδή τα κλασικά μέτρα ελέγχου που χρησιμοποιούμε, δεν είναι επαρκή, διότι υπάρχει το θέμα αρμοδιοτήτων του παράκτιου κράτους. Υπάρχουν κάποια όρια που έχουν σχέση με τις ε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και επίσης όλες αυτές οι δραστηριότητες συνεχώς μεταβάλλονται, γιατί δεν υπάρχει ένα διεθνές νεολόγιο. Έχουμε βέβαια σχέσεις με οργανισμούς Ενωμένων Εθνών και με περιφερειακούς οργανισμούς και μπορούμε να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα παγκόσμιο νεολόγιο για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εποπτεία. προς το παρόν παραμένω στο πεδίο της ευρωπαϊκής αλληλευτικής πολιτικής και μετά θα επεκταθώ και πέραν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Μας ενδιαφέρουν οι αλληλευτικές συμφωνίες και οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Είδαμε ποια είναι τα όρια αυτών των συμφωνιών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδίω ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτέ τι συμφωνίε και οι πολίτε του οποίου εκπροσωπείται ανησυχούν για αλληλευτικέ συμφωνίε με χώρε που δεν πληρούν τι ελάχιστε προποθέσει όσον αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα και τη διαφάνεια. Είναι θέματα που δημιουργούν ερωτηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα θεσμικά όργανα. Για το θέμα των εταιρικών σχέσεων, και θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Την περίπτωση ε, μιας αραβόφωνης χώρας που είχε ε, μια σύμβαση με την Κίνα που ήταν τουλάχιστον αδιαφανής ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς προτείνουμε πάρα πολύ διαφανή μέσα. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που συνάπτουν σκοτεινές συμφωνίες με άλλα συμβαλόμενα μέρη στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσης, στο πλαίσιο άλλων συμβάσεων, ίσως στο πλαίσιο της ΦΑΟ, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα μιας παγκόσμιας θέσπισης ε, ε, ε, αλληλευτικών συμφωνιών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί δεν θέλουμε μόνο εμείς να συνάπτουμε διαφανείς συμβάσεις και άλλες χώρες να συνάπτουν άλλες συμβάσεις αδιαφανείς. Θέλουμε η προσέγγιση μας έναντι του ελέγχου να είναι μια τέτοια προσέγγιση που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάλληλο, στο κατάλληλο πλαίσιο να θέσει σε εφαρμογή αυτά τα μέσα. Μπορεί να γίνει αυτό είτε διμερός, είτε στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης τη αλίας, όπω είναι στον Ατλαντικό ή η ΚΑΤ, και Ε, ξέρετε ότι υπάρχει και το πολύπλοκο θέμα των αποκλειστικών οικονομικών ε, ζωνών, ε, διότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί βάσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσα και για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στα ύδατα μια συμβαλόμενη χώρα ή μια παράκτητα χώρα θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε συμφωνίε. Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της ε, αυτούς τους περιορισμούς και προσπαθεί με αυτά τα οποία προτείνει ε, να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Κάτι άλλο που θα ήθελα τώρα να τονίσω είναι το θέμα της ε, βιωσιμότητας. Δηλαδή η κοινή ελευθερική πολιτική αποσκοπεί στη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Όταν εξετάσουμε την πρόσβαση στην αγορά, έχουμε τους σχετικούς κανόνες και διαπιστώνουμε ότι τα προϊόντα αλίας ε, έχουν ίδια μεταχείριση όπως τα εξαρτήματα αεροσκαφών ε, διότι είμαστε έξω από τον τομέα της γεωργίας. Η αλία ε, είναι ίδια διαχείριση όπως πριν από 4.000 χρόνια, από τότε που υπήρχε η Γεωργία και παλαιότερα. Μιλάμε για ιδιαίτερα ευάλωτα αγαθά που είναι περιβαλλοντικά αγαθά. γιατί να μην τροποποιήσουμε τους κανόνες πρόσβασης στην αγορά για τα λιευτικά προϊόντα έξω από το σύστημα των χωρών ΑΚΕ, του συστήματος, από το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων θεσπίζοντας συστήματα και βασίζοντας τα, τους τελωνιακούς δασμούς σε κανόνες βιωσιμότητας, δηλαδή ζητώντας από τις χώρες που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσουν κανόνες βιωσιμότητας και με βάση αυτούς τους κανόνες βιωσιμότητας να μπορούμε να δεχθούμε προϊόντα με ή χωρίς τελωνιακούς δασμούς. Είναι και αυτό λοιπόν ένα πιθανό μέσο καταπολέμησης της παράνομης αλίας. Ένα άλλο ερώτημα που μου κάνατε αφορά την διαθεσιμότητα των δεδομένων και ενδεχόμενες πιέσεις που θα μπορούσαν να ασκηθούν στον οργανισμό μας από τα κράτη-μέλη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση με νομικό τρόπο, γιατί ο κανονισμός της υπηρεσίας ελέγχου είναι ξεκάθαρος και το καταστατικό μας του 2005 αναφέρει σαφώς ότι ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της υπηρεσίας ελέγχου δεν λαμβάνει εντολές από τα κράτη-μέλη. Είναι μια ξεκάθαρη διάταξη και νομίζω ότι υπάρχει αυτονομία και η αίσθηση του καθήκοντος ε, που με διακρίνει δεν μπορεί να με αφήσει να μπω σε ε, ένα καθεστώς ελέγχου. και σας δηλώνω ότι θα υποβάλω την παρέτησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο ε, σε περίπτωση που ασκηθούν πιέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ε, υποχωρήσω σε τέτοιες πιέσεις. Ε, όσον αφορά τα δεδομένα, ο κ. Σκούν είπε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό δεδομένων. Όντω, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την συλλογή δεδομένων και την επεξεργασία τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία έχουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, σχέσεις εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας, μέσω πολλών κανονισμών, γιατί είχαμε τη μεταρρύθμιση του ελέγχου που αποτέλεσε μια κοπερνίκιο επανάσταση. Θέσπισε λοιπόν μαζί με τα κράτη-μέλη τις διατάξεις που αποκαλούμε σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Δηλαδή υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των αλλιευμάτων και των εκφορτώσεων μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Υλοποιείται τώρα αυτό το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου και θα συνεισφέρει στο να έχουμε μια πλήρη εικόνα των ποσοτήτων που αλλιεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των ποσοτήτων που εκφορτώνονται και των ποσοτήτων που πολλούνται. Προς το παρόν θα εφαρμοστεί για τα σκάφη πάνω από 12 μέτρα και οι πωλήσει, οι αγορές ε, ε, θα αφορούν ε, πάνω από 400.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τομέα και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι ζούμε σήμερα σε ένα κόσμο όπου όλοι οι οικονομικοί τομείς παρέχουν δεδομένα και το ίδιο πρέπει να κάνει και η αλληλεία. Ανακαλύπτουμε τα τελευταία χρόνια ποικίλε δραστηριότητε στο θαλάσσιο τομέα και η αλληλεία είναι μία από αυτέ τι δραστηριότητε. Προστασία των θαλασσίων χώρων, εγκατάσταση ανεμογεννητριών και άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στη συλλογή δεδομένων και η δραστηριότητα της αλίας θα συνεπάρχει με τις άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα του κ. Μπαρόζο για, το 2020 ε, συμπεριλαμβάνει μια σημαντική πτυχή που αφορά τις ε, βιώσιμες ενέργειες και η βιοπικιλότητα ε, είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του προγράμματος. Η αλληλεία λοιπόν και τα δεδομένα που μπορούμε εμείς να συγκεντρώσουμε μπορούν να συνεισφέρουν για τη βιώσιμη διαχείριση της θάλασσας. Σε ό,τι αφορά τώρα την πάνω μία αλληλεία στην Ισπανία ή σε άλλα κράτη-μέλη, νομίζω ότι πολλά κράτη-μέλη οι χάνοι έχουν ένα είδος ε, παραοικονομίας, ε, θα έλεγα, παράνομης τέλο πάντων αλληλευτικής ε, δραστηριότητας, αλλά νομίζω ότι αλλάζει η κατάσταση θα ελεγα παρανομης τελο παντων ληφτικης δραστηριοτητας αλλα νομιζω οτι αλλαζει η κατασταση επι του παρόντος. Όταν ξέρουμε πλέον τα δεδομένα μπορούμε να τα διασταυρώσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά είναι και νομικό το θέμα αυτό. Γιατί η Επιτροπή με τον κανονισμό για τον έλεγχο μπορεί να, δια... να, ε, να αναπτύξει έναν εκτελεστικό κανονισμό για τα επίγοντα μέτρα όταν η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ο κανονισμός αυτός που είναι ένας κανονισμός της επιτροπολογίας θα μπορούσε να δώσει στον οργανισμό, στην υπηρεσία, τη δυνατότητα να συζητήσει, να εξετάσει, να αντιμετωπίσει μια πολύπλοκη, ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση που έχει να κάνει με τα δεδομένα ή με την παράνομη αλία. Χρειάζεται όμως αυτός ο κανονισμός. Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη και τις σχέσεις εμπιστοσύνης, θα ήθελα να έχω τέτοιες σχέσεις και να μπορώ να καταλάβω ε, το πώς σκέφτεται για να δω και πώς ε, τελικά λειτουργεί η διοίκηση της αλίας σε κάθε κράτος μέλος. Και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις που μπορεί να είναι δυσχερείς ε, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Μου τέθηκε και ένα άλλο ερώτημα, το ερώτημα για το συντονισμό με τα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να σεβαστούμε τις ε, δυσκολίες που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι από το ένα κράτος στο άλλο, στο άλλο ε, διαφέρουν τα πράγματα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν ε, μέσα ελέγχου και συντονισμού πολύ επιτυχημένα παραδείγματο χάρη σχέδια κοινή ανάπτυξη. Νομίζω ότι η Κομισιόν μπορεί να συνεισφέρει, αλλά δεν είναι και απολύτω αναγκαίο αυτό, γιατί τα κράτη-μέλη νομίζω έχουν και τι ικανότητε ε, και τι αρμοδιότητε να διευθετήσουν μόνοι τους, ε, μόνα του τα πράγματα και η υπηρεσία είναι είδο διευκολυντή, δηλαδή φέρνει τα άτομα σε επαφή μεταξύ του. Μπορεί να συμμετέχει. Αλλά όχι τόσο γιατί τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ό,τι αφορά τους ε, πόρους είναι αυτά στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο. Μπορεί να έχουν μειωμένη αλληλεία, αλλά σίγουρα δυσκολεύονται να εφαρμόσουν το κοινοτικό και εκτιμένο και τις κοινοτικέ διατάξεις. Η υπηρεσία λοιπόν μπορεί να παρέμβει για να βοηθήσει αυτά τα κράτη να κάνουν μια διάγνωση της κατάστασης, να προσδιορίσουν τα πράγματα. Γι' αυτό και θέλω να έρθω ε, σε επαφή με όλα τα κράτη-μέλη, να προσδιορίσουν λοιπόν, να δουν σε ποιε περιοχέ θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση και σε ποιου τομεί, ό,τι αφορά την εκπαίδευση ή την ε, υλοποίηση των ε, σχεδίων ελέγχου. Και θέλουμε να έχουμε τα διάφορα σκάφη που μπορεί να φέρουν την Ισλανδική σημαία, αλλά να φέρουν και εμβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα συμμόρφωσης, να υπάρξει η εξέλιξη προς την υλοποίηση κοινών προτύπων από όλες τις χώρες και όλοι οι Ευρωπαίοι αλλοί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, να αντιμετωπίζονται δίκαια, ισότιμα και επίσης τα συστήματα καταστολής εφόσον αυτά ε, ενεργοποιηθούν να είναι και αυτά δίκαια και να εφαρμόζονται ισότιμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Μου τέθηκαν επίσης πολλά ερωτήματα για το σκουμπρί, ο πρόεδρος συγκεκριμένα, με ερώτηση για το σκουμπρί. Πράγματι, οι ποσοστώσεις, οι μονομερείς ποσοστώσεις, Ισλανδία, Φέροε και Ρωσία τώρα, πράγματι απαξιώνουν νομίζω τη διαχείριση της Αλίας στο Βόρειο Ατλαντικό που ήταν υποδειγματική μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δυσκολίες και ευτυχώς πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να διαπραγματευτεί μια δεκαετή συμφωνία ε, με την Ισλανδία για, το σκούμπρι με τη Νορβηγία, γιατί η Νορβηγία είναι εταίρος, ε, δεν είναι απέναντί μας σε αυτό το θέμα. Βέβαια, είναι κρίσιμη κατάσταση, γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν η Ισλανδία, η Ρωσία και η Φερόε δεν μειώσουν τα λεύματά τους, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή θα βρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση όπου είχαμε και με το προσφυγάκι, δηλαδή ε, κατάρρευση ε, των ΤΑΚ και πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ε, και πολλές δυσκολίες κυρίως για τους επαγγελματίες. Ή δεύτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Αλία θέλουμε να διατηρήσουμε τα λιεύματα και πρέπει οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι να καταβάλουν την προσπάθεια μειώνοντας τα λιεύματα με πολύ σημαντικές συνέπειε για την αλληλεία στην Ευρώπη. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη. Σε ορισμένα, ορισμένα κράτη-μέλη ε, υπάρχει σχεδόν ε, βιομηχανική αλία του σκουμπριού με πολύ μεγάλα σκάφη και ε, σχεδόν βιομηχανικού χαρακτήρα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε αλληλεία τεχνικού σχεδόν χαρακτήρα, όπου κάθε αλλιές αλλιέται μια μικρή ποσότητα. Και εδώ λοιπόν υπάρχει κάποια δυσκολία. Ε, δυστυχώς η υπηρεσία μας δεν μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα γιατί βρισκόμαστε λίγο έξω από την αποστολή μας. Η υπηρεσία μας όμως μπορεί να συμμετάσχει σε ελέγχους της κατάστασης στις Φερόες ή στην Ισλανδία με βάση στοιχεία που γνωρίζουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας υπόψη και αυτά τα οποία έχει δηλώσει η Ισλανδία, που κατά τη γνώμη μου είναι υπερεκτιμημένα. Στη συνέχεια, μπορεί να εγκαθιδρυθεί ένας διάλογος και να αποκατασταθούν οι σωστές σχέσεις με την Ισλανδία και τις Φερόες, ώστε να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα με τις χώρες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει κάποια μέτρα για τον έλεγχο των πελαγίων ε, ειδών και το σκουμπρί είναι ένα από αυτά τα είδη και θα υπάρχει ένα κοινό σχέδιο με τις χώρες αυτές για να μπορούμε να ελέγχουμε την αλία του σκουμπριού. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όπω αναφέρατε και εσεί, Πρόεδρε, υπήρχαν κάποια κράτη, και ανέφερε και η κυρία Αντρέα Μπαρέα, ε, κάποια κράτη που είχαν δυσκολίε στο παρελθόν και η Γαλλία είχε για τον ερυθρό τόνο δυσκολίε. Ε, Πολλέ χώρε έχουν δυσκολίε να τηρήσουν τα όσα έχουν θεσπιστεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουμε το πρόγραμμά μα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αηφόρο αλία. Όσον αφορά την Ισλανδία, Ε, φοβούμαι ότι εδώ έχουμε μία αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν δυνατότητες οικονομικών κυρώσεων, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ελπίζω να απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη που πήρα τόσο χρόνο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαβαρέ. Πληρέστατη απάντηση στις διάφορες ερωτήσεις που ετέθησαν από τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας στο μέλλον. Μπορείτε να μείνετε να ακούσετε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ίσως να σας ενδιαφέρει το επόμενο θέμα. Να δώσω ξανά στην Πρόεδρο, να παραδώσω ξανά την ε, Προεδρία στην Πρόεδρο. it's okay. Thank you. Ευχαριστώ. ευχαριστήσω τον κύριο Στίβενσον, διότι είχαμε μια συνέντευξη τύπου με τον ε, Πολωνό Υπουργό και με αντικατέστησε αυτό το διάστημα. Ζητώ συγγνώμη πάντως ε, από τον κύριο Σαβουρέ που δεν ήμουν παρούσα στην παρουσίαση που έκανε. Να σας πω επίσης ότι πρέπει να ε, ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον κύριο Ντεκόστερ και για το έργο του και για τις σχέσεις του με το Κοινοβούλιο και για την αφοσίωσή του, διότι πραγματικά ε, δρομολόγησε ε, και έστησε μια υπηρεσία ενώ ήταν αρκετά δύσκολες και πολύπλοκες οι συνθήκες. Τον κύριο Ντεκόστερ πραγματικά πρέπει να πω θα τον ευγνωμονούμε για όλα αυτά. Λυπούμε πραγματικά που αποχωρεί, ειλικρινά λυπούμε, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική φυσικά σχέση. Και βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εύχομαι κάθε επιτυχία και στον κύριο Σαβουρέ. Απλά θέλω να γραφεί στα πρακτικά η ευγνωμοσύνη που εκφράζουμε στον κύριο Ντεκόστερ για τις θυσίες του και για όλες τις προσπάθειές του για, ένα θέμα, για το οποίο ήταν βαθύς γνώστης. Μετά από όλα αυτά και περνάμε στο επόμενο σημείο της διάταξης. Πάλι 13. Α, τι γίνεται. 13ο σημείο λοιπόν. Τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση πολιετού σχεδίου αποκατάσταση του τόνου στο Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο με τον κύριο Ρωμέβα. Μα τα πει και ο κύριο Ρωμέβα. Από την Κομισιόν ποιον έχουμε εδώ, α, τον κύριο Ντενατέλα. Θέλετε να μιλήσετε πρώτος. Ή να δώσουμε το λόγο. Α, ωραία, ο κύριος Δενατέλα λοιπόν θα μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομο, προσπαθώντας να σας παρουσιάσω τα βασικά σημεία της πρότασης ε, τροποποίησης του κανονισμού του εφαρμοστικού που υθέτηκε το 2009 και έδινε συνέχεια στην έγκριση τέλους του 2008 του σχεδίου αποκατάστασης. Το Νοέμβριο του 2010 το ΙΚΑ τεθέτησε ένα σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου που συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία και όλες τις προόδους που προηγουμένως επετέφθησαν και αποφασίστηκαν ε, με νέα μέτρα επίσης όσον αφορά τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την εποπτεία τη γενική της εφαρμογής του σχεδίου αποκατάστασης. Ε, οι τροποποίησεις αφορούν επίσης το νέο πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται το σχέδιο αποκατάστασης που έχει σαν στόχο να καθορίσει και να δώσει στην Επιτροπή Εφαρμογή ένα ρόλο σημαντικότερο, όχι μόνο θα έλεγα εντό όσον αφορά τον εκτονιστέρων των έλεγχο τη συμμόρφωση των συμβαλωμένων μερών μετά την περίοδο αλλά να δώσει στην Επιτροπή Εφαρμογής του ΜΕΤΟ δυνατότητα πριν αλλιευτική περίοδο να γνωμοδοτεί επί του επίπεδου σεβασμού από πλευρά συμβαλωμένων μερών των διαφόρων διατάξεων του σχεδίου κυρίως κατά την προετοιμασία των αλληλευτικών σχεδίων, των σχεδίων ελέγχου και των σχεδίων ε, μείωσης της υπεραλύσης, του, υπερ, του δυναμικού. Εντάσσει λοιπόν τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνει τις, τα βασικά στοιχεία προηγουμένων αποφάσεων με νέες διατάξεις που θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίες ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις, το, τις δραστηριότητε δραστηριότητες στον τομέα και να αντιμετωπίσουμε και την εξέλιξη όσον αφορά τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται όσον αφορά ε, το που τοποθετείται ο τόνος ο αλλιευμένος από τα αλλιευτικά με Ανάμεσα στα νέα στοιχεία που αναφέρω το σχέδιο αποκατάστασης, να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία ήδη αναφέρθηκαν κυρίως εδώ, σε αυτή την Επιτροπή κατά παρελθόν, που εντοπίστηκαν ότι ήταν προβλήματα, αλλά χάρη στη συνεργασία με τα συμβαλόμενα μέρη καταφέραμε να φέρουμε βελτιώσεις και να δώσουμε τις δέσεις διευκρινήσεις. Ανάμεσα στα σημεία αυτά θα παραθέσω κάποια. Από αυτά θα ήθελα καταρχάς να αναφέρω το εξής για πρώτη φορά το σχέδιο αποκατάστασης θεσπίζει σαφέστατους κανόνες όσον αφορά την κοινή λειτουργία, κοινή αλληλεία, τα GFO αγγλιστή, και για πρώτη φορά ε, θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση στις κοινέ ελευτικές δραστηριότητε. Ε, θεσπίζει κάποιους ακριβέστερους ορισμούς περί των κοινών αυτών επιχειρήσεων και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των ορισμών κάναμε επιλογές επιλέξαμε να προτείνουμε καμία κοινή αλληλευτική δραστηριότητα να μην μπορεί να λαμβάνει χώρα μεταξύ ενό σκάφου με σημαία κάτω τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με σκάφου που έχει σημαία άλλου συμβαλωμένου μέρους Αυτό ήταν ένα στοιχείο που δημιούργησε πρόβλημα κατά το παρελθόν και για πρώτη φορά θα έλεγα διευκρινίζεται όσον αφορά τους κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση, τον έλεγχο και την εποπτεία, διότι έχουμε καθορίσει επίσης ποιες είναι οι υποχρεώσεις κυρίως όσον αφορά τη δήλωση των ε, αλλιευμάτων και αυτό αφορά και τα άλλα συμβαλόμενα μέρη βεβαίω, διότι η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο να απαγορεύσει αυτού του είδους τις αλλιευτικές δραστηριότητε ε, να καλύπτονται από σκάφη της Ευρωπαϊκής Και κάτι άλλο που θα αναφέρω, καλύτερη παρακολούθηση ε, όσον αφορά τις θέσεις ΒΜΕ των σκαφών. που κατά παρελθόν ήταν υποχρέωση που ίσχυε κατά τη διάρκεια της περίοδου της αλίας. Σε αυτό όμως το σχέδιο ανάκτησης, αποκατάστασης, η παρακολούθηση VMS γίνεται πριν από την περίοδο αλίας και μετά. Να αποφεύγουμε τη στιγμή όπου ε, η περίοδος αλίας, τα παρασυρώμενα δίχτυα, ξεκινάνε άλλα σκάφη για την ανοιχτή θάλασσα και δεν μπορούν να ανοιχνευτούν από το σύστημα VMS. Τρίτο στοιχείο. Όλο το σύστημα ελέγχου αναθεωρήθηκε και θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω όλος ιδιαίτερο το εξή. Έχουμε άρθρα εντελώς καινούρια για όλες τις επιχειρήσεις. Μεταφορά τόνου από αλλιευτικό σκάφος προς ρημουλικό σκάφος από το ρημουλικό σκάφος ε, προς τις ε, καλλιέργειες, εκεί τις, τους χώρους ανάπτυξης του, τόνου ε, και διαχείριση του ελέγχου εντός των κλοβών χωρίς να επισέθουμε τώρα σε λεπτομέρειες για τα νέα στοιχεία και τις νέες τεχνικές να διευκρινίσω ότι πρόκειται περί νέων κανόνων που ήδη μας επέτρεψαν καλύτερη εικόνα, καλύτερη γνώση του ακριβούς επίπεδου των αλλιευμάτων και του ακριβούς επίπεδου της βιομάζας στις διάφορες επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλληλευτική δραστηριότητα και τη θέση κλωβούς. αυτές ε, οι διατάξεις αποτελούν αντικείμενο διευκρινήσεων και στο πλαίσιο του ΙΚΑΤ. Και κλείνω τώρα αναφερόμενος σε αυτό που προανέφερα. Νέο είναι το πλαίσιο, νέα δεδομένα. Διευκρινίσαμε στο σχέδιο αποκατάστασης της υποχρεώσης όσον αφορά το reporting στο ΕΚΑΤ και στην Επιτροπή Εφαρμογής. Όπως θα διαπιστώσατε, η Επιτροπή, η εφαρμοστική, έλαβε νέες, ανέλαβε νέες ευθύνες, όπως προανέφερα. Φεβρουάριο του 2011, κατά διάρκεια τη συνεδριάσεω τη Επιτροπή Εφαρμογή, πριν από την περίοδο του 2011 τη Αλία, έπρεπε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουμε ένα σχέδιο αλλιευτικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώσεω του δυναμικού και σχέδιο ελέγχου και επιθεώρηση. Για την περίοδο 2011, αυτά τα σχέδια λοιπόν ενεκρίθησαν από την Επιτροπή και από την ΕΚΑΤ και αυτό μα επέτρεψε να αποφύγουμε πρόβλημα Όσον αφορά την λευτική δυνατότητα για το 2011, η ίδια επιχείρηση θα πρέπει να γίνει το ίδιο εγχείρημα και για την περίοδο 2012. Όχι το 2012, αλλά ήδη τώρα. Δηλαδή, όταν η Επιτροπή Συνεδρία τον Νοέμβριο του 2011, είναι μια δουλειά που θα χρειαστεί πάρα πολλέ προσπάθειε και από πλευρά κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα υπάρχουν διατάξει ακριβέστερε σε συγκρίση με το παρελθόν όσον αφορά τι υποχρεώσει που έχουν τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τα τρία ξεχωριστά σχέδια, καθώ και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να διαβιβάζει αυτά τα σχέδια από τη στιγμή που θα έχουν παραληφθεί από πλευρά κρατών μελών. Ιδού, κυρία Πρόεδρε, τι θέλω να πω για μια ακόμη φορά Αυτά αποτελούν προόδους που καμιά φορά είναι τεχνικής φύσεως, αλλά γενικά μας επιτρέπουν ήδη να έχουμε πιο σφαιρική εικόνα όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων και όχι μόνο των αληφτικών τιούτων, αλλά τη θέση εκλοβούς και τη μεταφορά ε, προς τη στεριά είναι ένα ε, σχέδιο αποκατάστασης που θέλει να ενισχύσει εν γέννη την επιθεώρηση και την παρατήρηση και την εποπτεία διότι ενισχύσαμε τα στοιχεία και τέλος έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε ένα ενίο έγγραφο που συμπεριλαμβάνει όλες τις διατάξεις του σχεδίου αποκατάστασης ενώ το κατά παρελθόν όταν υπήρχαν αλλαγές ήταν διαφορετικά τα πράγματα και σε ένα έγγραφο ξεχωριστό ε, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα ε, των ε, παρανόμων αλευμάτων εδώ έχουμε σφαιρική εποπτεία όσον αφορά τον έλεγχο και την επιθεώρηση και το, το σχέδιο αποκατάστασης. Κύριε Ρωμέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντενατέλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που είχαμε να μας εξηγήσετε εσείς το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βέβαια τα περιθώρια ελιγμών ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι μηδενικό υπό την έννοια ότι έχουν ληφθεί σε επίπεδο ή κάτι αποφάσει. Εκεί διαμορφώνονται οι απόψει και εκεί δίνονται οι μάχες. Ε, τέλος πάντων, Εμεί ω Κοινοβούλιο το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε όλα αυτά στο δικό μας επίπεδο, ε, στο δικό μας νομοθετικό επίπεδο. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση κατά το παρελθόν και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη συνεδρίαση της ΆΙΚΑΤ στην Κωνσταντινούπολη, που από ό,τι φαίνεται θα είναι μεταβατική. Δεν υπάρχει και κάποιο πολύ σημαντικό ζήτημα επιτάπητος. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε πτυχές οι οποίες θα συζητηθούν εκεί, που μπορεί να μην είναι αντικείμενο συζήτηση στη συγκεκριμένη αυτή πτυχή, αλλά στο τευρό το χρονοδιάγραμμα, το γεγονός πώς να το πω. Εμείς θα λάβουμε την απόφαση για την ε, μετάβαση λίγες μέρες πριν ή μετά την Κωνσταντινούπολη. Και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το κείμενο το οποίο θα έχει εγκριθεί στην Κωνσταντινούπολη στη δική μας απόφαση. Και ιστορικό, ήταν ιστορικός ο οργανικός διάλογος ε, που είχαμε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και σε ό,τι αφορά τι πράξη, για παράδειγμα, για το Κοινοβούλιο ήταν σαφέ. Εμεί προασπίζουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν αυτέ οι σε πράξη, αυτό το σύστημα, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να συζητηθούν ξανά κάποια θέματα, το ίδιο συμβαίνει και με το Συμβούλιο. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, υπάρχουν και πτυχές που θα προκαλέσουν συζητήσει. Παραδείγματο χάρη, κατάσταση στη Λιβύη, ότι υπάρχουν κάποια σκάφη που έφυγαν από ύδατα ή λιμάνια ευρωπαϊκά για να λιεύσουν στη Λιβύη και αυτά δεν τα ελέγχει κανένα γιατί ουσιαστικά πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ελέγχουμε τα ευρωπαϊκά σκάφη πάρα πολύ καλά, αλλά ελάχιστα ελέγχουμε του στόλου τρίτων χώρων. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα βέβαια ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα λεπτό ζήτημα ε, που έχει να κάνει με τα άλλα και εμείς δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή η καινοτομία, αυτό το νέο στοιχείο, ε, ε, οι κοινέ αποστολές αυτές, θα βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη πρόληψη αξιολόγηση τέτοιων καταστάσεων, που είναι και απειλητικέ. Η Ιαπωνία, επίσης ένα πρόβλημα, η κατάσταση στην Ιαπωνία. Δεν είναι τα ίδια τα πράγματα με πέρυσι και θα πρέπει να επανεξετάσουμε κάποιες συμφωνίες που έχουμε και να δούμε βέβαια ότι έχει αλλάξει και η οικονομική και εμπορική κατάσταση της Ιαπωνίας. Και αυτό επηρεάζει την όλη δραστηριότητα. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς η Ιαπωνία αλλά και οι προμηθευτές της Ιαπωνικής αγοράς να δούμε πώ θα αντιδράσουν. Αλλά να δούμε και την αντίδραση άλλων χωρών όπω τη Κίνα, για παράδειγμα. Να δούμε τι θα κάνουν οι Κινέζοι, πώς θα τοποθετηθούν σε αυτό το χώρο μείωση αλληλευτικού στόλου, έλεγχη, όλα αυτά πολύ καλά τα είπατε και νομίζω ότι παρόλα αυτά πράγματι υπάρχει σημαντική πρόοδος. Ένα μικρό ερώτημα ή μια μικρή παρατήρηση για αυτό το VCD. Το πρόβλημα είναι ο έλεγχος. Είναι δύσκολος ο έλεγχος, ακόμη και με την καλύτερη δυνατή βούληση από την διοίκηση. Ουσιαστικά εξαρτόμαστε από το πόσο αυστηρά ε, θα τηρούν ε, τις διαδικασίες οι αλλοίς. Δεν μπορούμε να έχουμε εγγύησεις Και κάποιες φορές τα δεδομένα που βλέπουμε δεν είναι απόλυτα ε, ορθά και γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Και έτσι δεν γίνεται κατανοητή ιδιαίτερα η κατάσταση ούτε η όλη διαχείριση με πάντω ευκαιρία και χαιρετούμε που είναι μαζί μα και ο κύριο Σαβουρέ, γιατί κατά το παρελθόν είχαμε ζητήσει πολλέ φορέ εδώ στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να έχουμε τι αξιολογήσει ε, τη υπηρεσία ελέγχου πριν πάμε στο ICAT, για να μπορούμε να λαμβάνουμε ε, αναλόγως και κάποιες αποφάσεις. Με τον κύριο Ντεκόστερ το είχαμε συζητήσει πολλές φορές και βελτιώσαμε Ε, όχι βέβαια κατά τρόπο απόλυτα ικανοποιητικό, αλλά τέλος πάντων βελτιώσαμε κάπως τα πράγματα. Χαίρομαι που είναι εδώ και λοιπόν και ο κύριος Σαβουρέ, ώστε επιτέλους ε, οριστικά να λύσουμε το πρόβλημα και να μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση πριν, να την έχουμε εκ των προτέρων, για να μπορούμε να κάνουμε τη δική μας ε, δουλειά ως πολιτική πιο σωστά. Θα αρχίσουμε τη δουλειά, θα δούμε μετά το καλοκαίρι πώ θα αποκρισταλωθούν όλα αυτά σε μια έκθεση που θα τη συζητήσουμε και με τι άλλε πολιτικέ ομάδε, με του άλλου συναδέλφου και βέβαια θα είμαστε ε, έτοιμοι να δούμε και τι άλλε αλλαγέ θα μπορούσαν να υπέρθουν μετά την συνεδρίαση τη ΆΙΚΑΤ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρο. Θα το συζητήσουμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρίασή μα ε, του Σεπτεμβρίου αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντενατέλα. Ε, και εδώ μπορώ να κηρύξω τη λήξη της σημερινής μας συνεδρίασης για το πρωί βέβαια, αλλά θα ξεκινήσουμε στις 3 με την παρουσία της Επιτρόπου κυρίας Δαμανά και σας ε, παρακαλώ να μελετήσετε τις προτάσεις. Πραγματικά και εγώ είμαστε όλοι νομίζω να τις διαβάσουμε.